Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de... Να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση που αφορά ένα θέμα μεγάλο ενδιαφέροντος για την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει να κάνει με τις ε, εταιρείε και τις, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σήμερα θα, θα γνωρίσουμε και θα αναλύσουμε το θέμα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται σε ένα πλαίσιο ε, που σχετίζεται με την αρπαγή γης. Ε, πέρα από αυτόν τον τίτλο υπάρχει μια πολύ σκληρή πραγματικότητα που απόψε θα αναλύσουμε μαζί με τους πρωταγωνιστές της. Πέρα από το να ευχαριστήσω καταρχάς τους εκπροσώπους των πρεσβειών, τους διπλωματικούς ε, εκπροσώπους που παρακολουθούν τη σημερινή συνεδρίαση, θα ήθελα να αποσαφηνίσω ότι στόχος αυτής της συνεδρίασης και της εργασίας μας δεν είναι να τονίσουμε στις κυβερνήσεις των τρίτων χωρών αλλά, το τι συμβαίνει, αλλά να συνειδητοποιήσουμε τις ευθύνε μας ως Ευρωπαίοι. Δηλαδή, είναι κατά τη γνώμη μας απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε όχι μόνο ως κοινωνίες αλλά και ως ε, επιχειρήσεις αλλά και δημόσιες ε, αρχές ε, της Ευρώπης το ρόλο που παίζουμε στις τέτοιες χώρες. Εμείς έχουμε αναλάβει υποχρεώσεις όσον αφορά την ανάπτυξη των λαών και θεωρούμε και ελπίζουμε και ότι οι κυβερνήσεις θα κάνουν το ίδιο. Ωστόσο, Είμαστε μέλη μιας ε, πολιτικής κοινότητας που έχει αρχές και αξίες εξαιρετικά στέρεες όσον αφορά την ανάγκη προστασίας των πιο αδύναμων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα γι' αυτό έχουν ε, θεσπιστεί, για να προστατεύουν τους πιο αδύναμους και γι' αυτό οι μεγάλοι όμιλοι οι τράπεζες, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο σύνολό τους θα πρέπει να δεσμεύονται ε, με ε, τον σεβασμό των αξιών που ανέκαθεν έχουν υπερασπιστεί οι Ευρωπαίοι πολίτες. Επιμένω λοιπόν ότι θα ακούσουμε σήμερα τους πρωταγωνιστές των ε, ιστοριών που οδήγησαν στην δίωξη ακόμα και στη δολοφενία ε, πολλών εξ αυτών όπως ε, η κυρία Κάθερες έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας την κόρη της την Βέρτα Θουνίχα Κάθερες που είναι η άξια κόρη, η άξια απόγονος της Βέρτα Κάθερες Η Μπέρτα Κάθερες εξακολουθεί να ζει χάρη στην κόρη της και Θέλουμε να, έτσι να επιβεβαιώσουμε ποιο είναι το καθήκον μας και ότι αυτή τη στιγμή η θέλησή μας για την τήρηση των στάνταρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος δεν μας νούν αρκετά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν χρειάζεται να θεσπιστούν δεσμευτικά μέσα, άμεση νομοθεσία, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και συγκεκριμένα οι ευρωπαϊκές εταιρείε να μην μπορούν ποτέ να ευνοήσουν αυτή τον τρόπο εξάλληψης γεών πληθυσμών χωρίς να προστατέψουν τις ζωές και τα συστήματα ζωής όλων αυτών των ανθρώπων. Είμαστε πεπισμένοι ότι είναι απαραίτητο να νομοθετήσουμε και να υποχρεώσουμε στο σεβασμό αυτών των αρχών. Θα σας παρουσιάσω τώρα τους ανθρώπους που θα πάρουν το λόγο σήμερα και που είναι άμεσα ε, ε, συνδεδεμένη με αυτές τους ε, αγώνες η κυρία Χάνα Σάρινεν που είναι σύμβουλος επενδύσεων στην γεωργική πολιτική στην Oxfam International και για την Ονδούρα όπως σας έλεγα Κοντά μας είναι η κόρη της Μπέρτα Κάθερες, η Μπέρτα Θουνίχα Κάθερες, που είναι μέλος της Κοπίν του Συμβολίου των Λαϊκών Οργανώσεων και των Οργανώσεων Αυτοχθόνων της ε, Ονδούρας που ήρθε ε, ώστε να μας μεταδώσει ε, από πρώτο χέρι ποια ήταν η δίωξη, η καταδίωξη που υπέστη η μητέρα της καθώς και η οργάνωσή της το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου στην ουσία. Διότι είχε λάβει άμεσα 33 φορές απειλές εναντίον της ζωής της μέχρι ότου δολοφονήθηκε τελικά. Ελπίζουμε πως θα έχουμε τη συνεργασία των αρχών της Ονδούρας. Ε, νομίζω πως είναι εδώ και οι εκπρόσωποι της διπλωματικής αντιπροσωπείας της Ονδούρας ώστε να ε, φωτιστεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη στην υπόθεση της Μπέρτας Κάθερες. Κοντά μας είναι επίσης η Λίντα Μπρικουζεν που είναι επικεφαλής ε, το επενδυτικού τμήματος της Ολλανδικής Τράπεζας Αναπτύξεως που ε, ε, έχει επενδύσει στο σχέδιο Άγουα Θάρκα και που παρακολούθησε όλες τις ε, συγκρούσεις και τις αψημαχίες με την Κοπίν και που πριν από λίγες εβδομάδες απέσυρε τη χρηματοδότηση για αυτό το έργο. Έχαστη για την Κολομβία έχουμε τον ε, πατέρα Αλβέρτο Φράγκο που είναι μέρος της ε, Διεκκλησιαστικής Επιτροπής Δικαιοσύνης και Ειρήνης ε, της χώρας και επίσης θα δούμε και άλλη μια περίπτωση στη Λιβυρία, άλλο μέρος του κόσμου, με τον κύριο Άλλη Κάμπα από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης της χώρας του. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε σήμερα και χωρίς άλλη καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στην κυρία Χάνα Σάρινεν για την πρώτη γενική εισήγηση. Παρακαλώ. Good afternoon and thank you, um, Chair. Καλησπέρα σας ε, και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες ε, και κύριοι βουλευτές. Εργάζομαι στην Oxfam, βρίσκομαι εδώ πέρα στο γραφείο των Βρυξελών και σήμερα θα σας δώσω μια εικόνα των σχέσεων μεταξύ διεθνών οικονομικών ε, οργανισμών και αυτών των δικαιωμάτων, συγκεκριμένα της αρπαγής γης. Πρώτα απ' όλα, ποια, ποιοι είναι οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Είναι διάφοροι φορείς, έχουν διαφορετικές έντολες και ορισμούς. Δεν είναι πάντα ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι οι λεγόμενοι οργανισμοί αναπτυξιακής χρηματοδότηση με εντολή να επενδύσουν σε αναψώμενες χώρες για να δημιουργήσουν ανάπτυξη και ταυτόχρονα να έχουν και κάποιο οικονομικό αποτέλεσμα. Παραδείγματο χάρη η Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΦΗ των οργανισμών αυτών ε, αριθμεί 15 μέλη όπως το FMO, το KFV, το γερμανικό η Βελγική Οργάνωση Αναπτυξιακής Βοήθειας κτλ. Επίσης υπάρχουν οι πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, οι οποίες παρέχουν οικονομική στήριξη και συμβουλές για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εδώ πέρα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα, το παγκόσμιο, το περιφερειακό και το υποπεριφερειακό. Π.χ. στο παγκόσμιο επίπεδο έχουμε την Παγκόσμια Τράπεζα και τη νέα αναπτυξιακή τράπεζα που συναισθήθη πρόσφατα από τις χώρες BRICS, τις λεγόμενες. Μετά στο περιφερειακό επίπεδο υπάρχει η Αφρικανική, η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ασιατική Τράπεζα Υποδομών, η Αμερικανική Τράπεζα ανάπτυξη και μετά υπάρχει η ΚΑΜΠΕΗ στην Κεντρική Αμερική, η Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανατολικής Αφρικής. Λίγα παραδείγματα είναι αυτά. Υπάρχουν πολλά τέτοια, πολλοί τέτοιοι οργανισμοί. Κάποια από αυτά έχουν ξεκάθαρη εντολή να εξαλείψουν την φτώχεια, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η οι άλλες αναπτυξιακέ τράπεζε, ενώ άλλε έχουν ε, ρόλο την πρόθεση της οικονομικής ανάπτυξης ε, και τη ανθρώπινης ανάπτυξης στις ε, περιοχές τους η καθεμία. Ο ρόλος των διεθνών αυτών οργανισμών αυξάνεται συνεχώς. Παραδείγματος χάρη πέρσι στο σχετικό σεμινάριο τονίστηκε ο ρόλος που μπορεί να παίξουν ε, στο να στηρίξουν την αηφόρο ανάπτυξη εφαρμόζοντας και τους στόχους ε, της, ε, τους αναπτυξιακούς και με την παροχή εμπειρογνωμοσύνης. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο μεγαλύτερος τέτοιος οργανισμός. Για να σας δώσω μια ιδέα του ισολογισμού της, μιλάμε για 540 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, τα νούμερα του 2014 είναι αυτά και έχουν αυξηθεί κιόλα. Και τα 15 μέλη της ε, ΔΕ έχουν 30 δισεκατομμύρια ευρώ έναν επενδυτικό φάκελο και επενδύουν σε πάρα πολλά έργα παγκοσμίω και πολλές, ε, πολλά κράτη, η Ολλανδία, η Φιλανδία αφιερώνουν μεγάλο κομμάτι στην αναπτυξιακή βοήθεια που περνάει μέσα από τα δικά τους θεσμικά όργανα. Οι περισσότερες από τις λειτουργίες είναι επικεντρωμένες στις οικονομικές υποδομές, ε, π.χ. σε δρόμους, αεροδρόμια, υποδομές ενέργειας, φράγματα παραδείγματος χάρη. Και τα έργα αυτά έχουν ε, δυνητικά μια επίπτωση στη χρήση γης και συχνά μπορεί να καταλήγουν σε εκτοπισμούς ε, εντόπιων κοινοτήτων. Οπότε όταν μιλάμε για τα δικαιώματα της γης υπάρχει ένα μεγάλο κενό παγκοσμίω. Μέχρι έως και 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίω εξαρτώνται από την γη και τους φυσικούς πόρους για να επιβιώσουν. Ε, ένα τρίτο του πληθυσμού του παγκοσμίου. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αγρότες, άντρες και γυναίκες, ψαράδες που αντλούν δηλαδή άμεσα τα προστοζήνα από τη χρήση γης και φυσικών πόρων. Μπορεί να είναι και αυτόχθονες ε, πληθυσμοί ή άλλες ε, τοπικές κοινότητες. Κατέχουν περιοχές που καλύπτουν πάνω από το 50% της ε, έκτασης του πλανήτη, όμως νομικά κατέχουν μόνο το 10%. Και αυτό είναι το κενό ακριβώς που υπάρχει. Καταλαμβάνουν, όπως είπα, 50% της ε, επιφάνειας ε, του πλανήτη, αλλά νομίμως κατέχουν μόλις το 10%. Και το υπόλοιπο είναι με διάφορα καθεστώτα χρησικτησίας ε, και άλλα τέτοια τα οποία σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ευάλωτοι σε πιο ισχυρούς και είναι βεβαίως στο έλεος των αρπαγών γης. Οι αριθμοί είναι από μια έκθεση ονόματι Common Grounds που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τον δικό μας οργανισμό και άλλους στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που κάνουμε για να κλείσει αυτό το κενό έτσι ώστε οι αυτόφανες ε, λαοί και οι τοπικές κοινότητες που χρησιμοποιούν αυτούς τους πόρους ε, εθιμικά να αναγνωριστούν από την εθνική τους νομοθεσία. Μπορείτε να βρείτε αντίγραφα στην είσοδο. Έχει υπάρξει κάποια πρόοδος προσφάτως στο θέμα αυτό, αλλά πολλά πρέπει ακόμα να γίνουν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να περάσουν καλύτεροι οι νόμοι, νέοι νόμοι και βεβαίως υπάρχουν ακόμα πολλά κενά για να είναι αποτελεσματικοί αυτοί οι νόμοι, να εφαρμόζονται. γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρουν ε, τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Ε, πρώτα απ' όλα είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θέμα αξιοπρέπειας, ε, σεβασμού για τις κοινότητες αυτές. Είναι θέμα ανάπτυξης επίσης. Παραδείγματο χάρη στην Ινδία γύρω στο 50% των οικοκυριών της υπαίθρου αντλούν τα προστοζήνα απευθεία από κοινόχρηστε εκτάσεις. Στην Αφρική επίσης 90% της γή της υπαίθρου στην Αφρική δεν είναι καταγεγραμμένη, κατά το οποίο συνδέεται άμεσα με τα υψηλά ποσοστά φτώχειας. Επίσης, ε, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στην γη ε, έχουν ένα ρόλο να παίξουν στην καταπολέμηση της ε, κλιματικής ε, αλλαγής. Πρόκειται πραγματικά για πάρα πολύ σημαντικά σημεία για την βιοπικιλότητα και εκεί πέρα βρίσκεται 80% της βιοπικιλότητας του πλανήτη. Και τέλος, έχουν σημασία, όπως είπαμε, και για καλύτερες επενδύσεις. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι οι συγκρούσεις για τη γη αυξάνονται Υπάρχει επίσης ένα οικονομικό τίμημα των συγκρούσεων αυτών. Το Πανεπιστήμιο της Queensland εκτιμά πως οι συγκρόσεις αυτές είναι περίπου το 50% του οικονομικού κινδύνου των επενδύσεων στον εξορρυκτικό κλάδο. Μια άλλη εκτίμηση λέει πως ε, αν δεν υπάρχουν ε, ασφαλή τέτοια δικαιώματα μπορεί να αυξηθεί και να ενιαπλασιαστεί ακόμα το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ενώ λοιπόν το κενό αυτό δεν ε, κλείνει, βλέπουμε περιπτώσεις παραβιάσεων των δικαιωμάτων. Να σας αναφέρω κάποια. Π.χ. υπάρχει μια επένδυση της International Finance Corporation στην Dragon Capital που βασίζεται στο, με έδρα το Βιετνάμ και με πελάτη την ε, HAGL με παραχώρηση χρήσης γης 50.000 εκταρίων στην Καμπότζη και στο Λάος οι οποίες ε, καλλιεργούνται αυτή τη στιγμή από άλλους ε, και βεβαίως αυτό θα είναι καταστροφικό για το αν θα μπορέσουν να επιζήσουν. Επίση υπάρχει πάλι από τον ίδιο οργανισμό μια επένδυση 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ταμείο Υποδομών της ε, Ινδίας που οδήγησε μια καταγγελία για το ότι επηρεάζονται αρνητικά 5.000 άτομα. Στην Ονδούρα υπάρχει περίπτωση του FMO και της IFC που εμπλέκονται στην Banco Ficoza και την επιχείρηση Corporation Dinant όπου πλέον ε, είχαμε φτάσει και σε δολοφονίες. κάποια παραδείγματα αυτά συγκρούσεων που λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Ένα λεπτό έχετε ακόμα. Συχνά το πρόβλημα είναι πως οι κοινότητες και τα άτομα που υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους ε, θεωρείται ότι προκαλούν ε, φασαρίες, ότι είναι ταραχοποιοί, τους απειλούν. Γύρω στα χίλια τέτοια άτομα έχουν δολοφονηθεί από το 2002. Αυτά έχουν καταγραφεί, έχουμε πάλι όπως σας είπα περισσότερες πληροφορίες στην είσοδο της ε, αίθουσας. Συγκεκριμένα τώρα για την ε, περίπτωση εδώ της Άγουας Άρκα που μας απασχολεί. Καταδικάζουμε δολοφονία της Κάρσερες ε, και της Αταγκαρσίας. Ζητήσαμε από τις αρχές να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη έρευνα υπό την εποπτεία της Αμερικανικής Επιτροπής ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητάμε από την κυβέρνηση της χώρας να προστατεύσει όσοι υπερασπίζονται τα δικαιώματα στους φυσικούς πόρους ε, και βεβαίως να βελτιώσουν την αξιολόγηση του κινδύνου και τις δικλείδες ασφαλείας για να αποφευθούν τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν επενδύουν ε, πολυμερείς οργανισμοί μέσω ενδιαμέσων. Συχνά δηλαδή δεν δίνεται το βάνιο η επιχορήγηση απευθείας, αλλά μέχρι και 70% των ε, δανείων πηγαίνουν μέσω ενδιαμέσων και στη διαδικασία αυτή υπάρχει ψηλός κίνδυνος ε, να υπάρχει αδιαφάνεια όσον αφορά την πληροφόρηση και οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές δικλίδες που θα έπρεπε να υπάρχουν και για τις οποίες έχουν δεσμευτεί οι διεθνείς οργανισμοί να μην γίνονται σεβαστοί. Τώρα, ποιε είναι οι συστάσει μα ε, προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρξουν πολιτικέ οι οποίε θα αναγνωρίζουν και θα προστατεύουν τα δικαιώματα των κοινοτήτων στη χρήση γη σε όλα τα έργα και τι λειτουργίε και να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει επαρκής και στοχευμένη αναπτυξιακή βοήθεια για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα στην γη και να υπάρξει βεβαίως και νομική ενδυνάμωση και δυνατότητα προσφυγής των κοινοτήτων να υπάρξει επίσης ε, μια, να υπάρχει πρώτερη συνένωση των ε, κοινοτήτων αυτών και θα πρέπει βεβαίως να σέβονται και τον κώδικα ΕΦΠΙΚ και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πρωτοπορεί την εφαρμογή των εθελοντικών κατευθυντήριων γραμμών που ε, προτείνουμε για όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα και τις ε, επιχειρήσης. Θα πρέπει επίσης ε, να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί προσφυγής ε, και λόγοδοσίας όσον αφορά τους ιδιώτες επενδυτές και τις επιχειρήσεις οι οποίες προμηθεύονται άγαθα και ζητάμε επίσης να υπάρξει μια δέσμευση για να μην προκαλείται ζημία μέσω του εμπορίου, επενδύσεων ή άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηριχθούν οι αυτόχθονες ε, πληθυσμοί και οι τοπικές κοινότητες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, λυπάμαι που είμαι κάπως αυστηρή με το χρόνο, αλλά δεν έχουμε τόσο πολύ στη διάθεσή μας. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Πέρτα του Νίχα Κάθρης και μετά η Ολλανδική Επενδυτική Τράπεζα που είναι μαζί μας ε, ώστε να δούμε πιο σφαιρικά την υπόθεση. Παρακαλώ. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, ονομάζομαι Μπέρτα Σουνίχα Κάθερες και το 2 Μαρτίου η μητέρα μου Μπέρτα Κάθερες δολοφονήθηκε δύο μέρες πριν από τα γενέθλιά της, ε, τα 45 γενέθλιά της. Ο θάνατός της είναι απώλεια για ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και ακούστηκε ε, αυτός ο θρήνος ε, παντού. Ε, στις 2 Μαρτίου ο κόσμος έμεινε χωρίς μια υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποφιέρωσε όλη της την ενέργεια στο να κάνει πραγματικότητα τις διεθνείς δεσμεύσεις για την υπεράσπιση των ποταμών, των ε, λιβαδιών, των αρχαίγωνων ε, ε, εδαφών στην αξιοπρεπή ζωή ενάντια στη μοντέλα στιγμής εκμετάλλευσης και υπέρ των δικαιωμάτων κυρίως των γυναικών. Στην Ονδούρα έγινε ένα πραξικόπημα το οποίο αλλάζει εντελώς την πραγματικότητα της χώρας μας. Το 40% της επικράτειας δίνεται σε εκχωρήσεις για την εγκατάσταση projects υδροελεκτρικών και εξορυκτικών εφαρμόζουν σε ολόκληρη την Ονδούρα αυτό ε, το σύστημα, ωστόσο συγκεντρώνεται στις, ε, στην επικράτεια των ε, αυτοχθόνων, οι οποίοι ζουν σε αρμονία με την φύση και συντηρούν τη φύση. Δίνονται λοιπόν στις επιχειρήσεις που τις μετατρέπουν αυτές τις περιοχές σε εμπορεύματα. Σύμφωνα με στοιχεία, ο αριθμός των υπερασπιστών που διώκονται ποινικά έχει αυξηθεί και φτάνει μάλιστα τις 3 1.850 υποθέσεις ε, ποινικοποίησης από το 2009 μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν δολοφονήθηκαν 15 υπερασπιστές και υπερασπίστριες των φυσικών πόρων και των ε, εδαφών που έπρεπε να προστατεύονται κανονικά. Σύμφωνα με την έκθεση της Global Witness στην Ονδούρα, υπάρχει ο μεγαλύτερος, ε, διαπράτεται ο μεγαλύτερος αριθμός δολοφονιών κατά κεφαλήν όσον αφορά τους υπερασπιστές ε, των εδαφών και του περιβάλλοντος στον κόσμο. Το 2010 μέχρι το 2015 τουλάχιστον 109 άνθρωποι έχασαν έτσι τη ζωή τους, δολοφονήθηκαν επειδή υπεράσπιζαν το περιβάλλον και τις αγροτικές ε, περιοχές. Η μαμά μου ήταν ένας άνθρωπος που διαρκώς απειλεί το επειδή υποστήριζε τις πεπιθήσεις της, υπερασπίζοντας ε, τα, δικαιώμα, τα δικαιώματα του αυτόχθωνα λαού, των Λέγκα. Από το 2013, όταν ξεκινάει η εγκατάσταση του υδροελεκτρικού project Agua Tharca, ε, που κατασκευάζεται από την ανώνυμη εταιρεία DESA της Ονδούρας, αυξάνονται οι απειλές και εντατικοποιούνται ε, ε, ε, δέχτηκε εκφοβισμό, απειλήθηκε με θάνατο και δύο φορές δέχτηκε επιθέσεις και επίσης διώχθηκε ποινικά στα δικαστήρια της Σονδούρα. Η ποινικοποίηση της και της οργάνωσής της που αγωνίζεται εδώ και 23 χρόνια ήταν μια τακτική πρακτική της εταιρείας, μια στρατηγική για να την αναγκάσει να, μάλλον, να, να, να θεσμοθετήσει, μάλλον να καταστήσει παράνομη την εργασία της και την εργασία της Σκοπίν. Η εταιρεία λοιπόν προσπαθεί τώρα να αρνηθεί τις ευθύνες της για αυτή την δολοφονία. Η μητέρα μου έλαβε ε, ε, δημοσία 33 απειλές που σχετίζονται με την εταιρεία και αυτά ήταν γνωστά στο κράτος. Η αδειοδότηση στην ΤΕΣΑ δόθηκε, σε αυτή την εταιρεία δηλαδή εκμετάλλευσης, δόθηκε στη διάρκεια του πραξικοπήματος και επίσης δεν έγινε σεβαστή η διαδικασία της πρώτερης ενημέρωσης ελεύθερη, της ελεύθερης πρώτερης ενημέρωσης και συνένεσης, ο κώδικας ε, ΦΠΙΚ. Ε, δεν σταμάτησε η κατασκευή των εγκαταστάσεων παρότι θεωρήθηκε η βασική πηγή των απειλών κατά τη ζωή της μητέρας μου. Αυτό το σχέδιο της, ε, του θανάτου έχει υλοποιηθεί με τη συνεργασία συνεργασία διεθνών τραπεζών όπως είναι η Ολλανδική Αναπτυξιακή Τράπεζα και άλλες εταιρείε, όπως η Siemens. Και εγώ ρωτώ, αυτά τα project που, όπου υπάρχει σαφής σύγκρουση ε, πρέπει να συνεχίζουν να κατασκευάζονται εάν αν δεν υπάρχει σύγκρουση, γιατί υπάρχουν νεκροί. Γιατί είναι νεκροί η Πάολα Κονσάλες, γιατί ο Βίλιαμ και ο Ροντρίγκε είναι νεκροί γιατί ένας ε, στρατιωτικός ο οποίος ε, φιλούσε το καρτέλ της ΔΕΣΑ κατηγορήθηκε για την δολοφονία του Τόμας Γκαρσία, γιατί είναι νεκρή η μητέρα μου γιατί οι χρηματοδοτικές τράπεζες εμπιστεύονται ε, και αναλαμβάνουν την ε, ηθική εξουσία ώστε να αποφασίζουν ποιοι είναι οι αυτόχθονες και ποιοι δεν είναι. Γιατί οι τράπεζες μπορούν να καταπατούν αρχές, αξίες ή μήπως τα ιδιωτικά συμφέροντα τα οικονομικά συμφέροντα αξίζουν περισσότερο από τις ζωές των αυτοχθόνων λαών. Αν έτσι είναι, έχουμε επανέλθει στην απεικιοκρατική εποχή. Αυτό που εμείς πιστεύουμε είναι πως ε, αυτή είναι μια ευκαιρία για να δημιουργηθούν δεσμευτικοί κανονισμοί για τους ε, διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους ε, έργα, για να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες των πράξεών τους. Γι' αυτό και ζητάμε την οριστική ε, ανάκληση των κονδυλίων που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία ε, DESA. Αυτά τα έργα του θανάτου δεν μπορούν να συνεχίζουν να κατασκευάζονται και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος αυτών των έργων δεν μετράται, με κιλοβάτ αλλά με αριθμό νεκρών. Η κυβέρνηση της Ονδούρα δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων των εξωτερικών βιομηχανιών. Σήμερα, 48 μέρες από τη δολοφονία της, η κυβέρνηση της Ονδούρα επανέλαβε σε διάφορες ευκαιρίες ε, την ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μάλλον κατηγορείται στα διεθνή βήματα για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αρνείται να ξεκινήσει διαδικασία έρευνας και ανακρίσεων για τη δολοφονία της μητέρας μου. Δεν εμπιστευόμαστε λοιπόν ε, θεσμούς που έχουν τοποθετηθεί υπέρ μιας επιχείρησης που συμμετείχε στην δίωξη, στην καταδίωξη δίωξη, στην εγκληματοποίηση, στην ποινικοποίηση τη δράση της, και τέλο τη δολοφονία τη μητέρα μου. Γι' αυτό και απαιτούμε τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής Έρεύνη μέσω της ε, Αμερικανικής ε, Επιτροπής ε, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ήδη έχει δείξει διαθεσιμότητα για να συστήσει μια τέτοια επιτροπή. Θέλουμε να πούμε ότι Εάν στην Οδούρα ένας άνθρωπος του μεγέθους της μητέρας μου δολοφονήθηκε, δεν ξέρουμε τι περιμένουν τους υπόλοιπους υπερασπιστές και υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που τοποθετείται σταθερά υπέρ της δικαιοσύνης και της προσπάθειας να σταματήσει ο θάνατος, η βία και η ατιμορρησία κάνουμε έκκληση να στηρίξετε αυτά τα αιτήματά μας και να συνεχίσετε αυτές τις χειρονομίες αλληλεγγύης στην αναζήτηση της δικαιοσύνης. Σήμερα, 48 μέρες από τη δολοφονία της, υποστηρίζουμε ότι έκαναν λάθος ε, η δολοφόνη. Η μητέρα μου ήταν ο φύλακας των ποταμιών. Ήταν μια δάμαστη γυναίκα και έχει υπερβεί το θάνατο. Δεν ε, πέθανε, πολλαπλασιάστηκε στον αγώνα κατά του θανάτου. Στον αγώνα υπέρ της ζωής. Γιατί τώρα όλοι είμαστε ε, τα φερέφωνα της. Ολόκληρος ο λαός ε, του Λέγκα της Ονδούρα. Δεν θα επιτρέψουμε αυτό το έγκλημα να περάσει ατιμόρυτη, αλλά θα πρέπει να αντίθετα να διερευνηθεί. Η αγάπη είναι ο πιο δυνατός κινητήρα στην αναζήτηση της δικαιοσύνης, μιας βαθιάς και πραγματικής δικαιοσύνης. Και κλείνω αυτή μου την παρέμβαση με τα λόγια της μητέρας μου. Ξύπνα ανθρωπότητα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, Μπέρτα. Τώρα το λόγο θα πάρει η κυρία Λίντα Μπροκούζεν, μάλλον λάθος ε, το πρόφερα, που είναι εκπρόσωπος της ε, Ολλανδικής Τράπεζας Ανάπτυξης. Παρακαλώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή οικογένεια και φίλοι της Κασιέρας, αγαπητοί εκπρόσωποι άλλων οργανισμών, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου προσφέρετε να απευθυνθώ σε αυτή την υποεπιτροπή Αρχικά θα ήθελα να δηλώσω ότι ειλικρινά λυπάμαι ε, για τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν ε, στο θάνατο, στη δολοφονία της κυρίας Κασέρες, τα συλληπιτήριά μου στους ε, φίλους και συγγενείς που μένουν πίσω. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τον πόνο που βιώνεται. καλέσαμε την κυβέρνηση της Ονδούρας να κάνει μια αναλυτική έρευνα ε, και να, ε, ε, να καλέσει σε λογοδοσία τους υπεύθυνους συναντηθήκαμε ε, με εκπροσώπους της κυβέρνησης για να υπάρξει μια έρευνα και να ε, υπάρξει μια βελτίωση της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ονδούρα. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η ελευθερία λόγου για αυτούς οι οποίοι υπερασπίζονται τα δικαιώματα ανθρώπων είναι υψής της σημασίας για εμένα αλλά και για όλους. Κάθε ε, άτομο θα πρέπει να νιώθει ασφαλές όταν υπερασπίζεται τη θέση του η FMO λοιπόν καταδικάζει οποιαδήποτε βία απέναντι σε αυτές τις ομάδες αλλά και σε ανθρώπους. Όντας ερευνήτρια για αρκετά χρόνια στην Ονδούρα μέσω ε, της ε, εταιρείας μας θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να βελτιώσουν τις ζωές τους. Προτεραιότητά μας είναι να ε, δεσμευτούμε με όλες τις πλευρές, ε, τόσο τις, αυτές που είναι υπέρ ημών όσο και τις κατά, μέσω ε, διαβουλεύσεων Θέλουμε οι επενδύσεις μας να συνεισφέρουν θετικά όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Τώρα όσον αφορά ε, το ε, ζήτημα ε, της δέουσας επιμέλειας, αυτό είναι κάτι το οποίο προσέχουμε ιδιαιτέρως. Ακολουθούμε πρότυπα αριστείας, υπερασπιζόμαστε την υπευθυνότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επίσης υποστηρίζουμε το ε, πλαίσιο του ΟΗΕ για την προστασία και το σεβασμό. Αυτή τη στιγμή κανονικά θα σας έδειχνα μια μικρή ε, ταινία σχετικά με το πρόγραμμα αό για να δείτε ε, τι δουλειά έχουμε κάνει ακριβώς και πόσο ακούσαμε ε, του ντόπιου πληθυσμό και το πόσο σημασία δίνουμε ε, στην ελεύθερη ε, πρώτερη και ε, έγκυρη συνένεση. Βέβαια, λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν λειτουργεί. Το link όμως για την ταινία έχει αποσταλεί σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Σας προσκαλώ λοιπόν να δείτε τη συγκεκριμένη ταινία διότι ε, μέσα ε, σε σύντομο χρονικό διάστημα δείχνει μια γενικότερη εικόνα του ε, προγράμματος καθώς επίσης και το έργο το οποίο έχουμε κάνει ως τώρα. Ακούσαμε προσεκτικά τους ντόπιου πληθυσμούς και λάβαμε δράσεις ε, ούτως ώστε να αλλάξουμε το πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτούμε προς ένα διαφορετικό πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τα όσα μας ήπιαν οι ντόπιοι πληθυσμοί και διασφαλίζοντας ότι ακούσαμε τις ανησυχίες τους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ταυτόχρονα η FMO ανησυχεί για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ονδούρα και υποστηρίζει ιδιαιτέρως ε, την ε, ε, κοινή πρόταση για υιοθέτηση μιας απόφασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεδομένή τη παρούσα κατάσταση και τη συνεχιζόμενης ε, βία αποφασίσαμε να σταματήσουμε τις δραστηριότητες μα στη χώρα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το FMO δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε νέα προγράμματα ή δεσμεύσει στην Ονδούρα. Δεν πρόκειται να υπάρξουν περαιτέρω πληρωμές ε, για το σχέδιο αυτό και ε, θα γίνουν περαιτέρω έρευνε όσον αφορά τις την υπάρχουσα κατάσταση, το αν θα αποχωρήσουμε ε, από το πρόγραμμα είναι ένα φυσιολογικό ερώτημα και είναι ερώτημα το οποίο θα θέτουμε και στους εαυτούς μας θεωρούμε ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στις διαδηλώσεις, ε, στις διαδηλώσεις ε, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ε, τα όσα έχουν πει λοιπόν τα ακούσαμε, ενώ υπάρχουν και ανεξάρτητοι σύμβουλοι που μας ενημέρωσαν για αυτό. Παρ' όλα αυτά οι έρευνες συνεχίζονται πάνω σε αυτό και γι' αυτό το λόγο οργανώνουμε μια αποστολή προς την Ονδούρα και καλούμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλό μας να μεταβεί εκεί πέρα για να ε, παρακολουθήσει από κοντά την κατάσταση και αυτό θα γίνει μόλις το, το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας. Ως Αναπτυξιακή Τράπεζα λειτουργούμε σε αναπτυσσόμενους χώρους με πολύπλοκα περιβάλλοντα και γι' αυτό το λόγο για εμάς ε, αποτελεί υψίστη προτεραιότητα να συμμετάσχουν όλοι οι παράγοντες στη διαδικασία, να έχουμε διαβούλευση και διάλογο και να μην αφαιρέσουμε ε, την αποζημίωση από ανθρώπους που το δικαιούνται και να διασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις συνεισφέρουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ε, βοηθούν στην καταπολέμηση κατά της φτώχειας. Επίσης, έχουμε έναν μηχανισμό αποζημιώσεων που αναφέρθηκε στην αρχή και ο οποίος είναι ανοιχτός οποιοδήποτε θέλει να διαμαρτυρηθεί για τα έργα μας. Εν τέλει είμαι πεπισμένη ότι τα ε, συμφέροντά μας είναι ισορροπημένα. Όλοι θέλουμε να εξαλείψουμε τη φτώχεια, θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και μια καλύτερη ζωή για το λαό της Ονδούρας. Γι' αυτό το λόγο το FMO καλωσορίζει ε, τις πληροφορίες ε, από εξωτερικούς παράγοντες όπως η ΜΚΟ, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα έργα μας γίνονται σωστά. Έχουμε μια συνάντηση στην Ολλανδία την επόμενη εβδομάδα με την κυρία Κασέρες, καθώς επίσης και με μέλη της Κοπίν, μια ΜΚΟ της Ονδούρας, όπου θα ακούσουμε ε, τις ανησυχίες τους καλούμε όλους τους παράγοντες ε, να συζητήσουν μαζί μας σε έναν ανοιχτό και επικοδομητικό διάλογο και καλωσορίζουμε οποιαδήποτε πρόταση για να βελτιωθούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Τελικά να αντιμετωπίσετε και να ξεκαθαρίσετε την κατάσταση. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, πατέρα Αλβέρτο Φράγκο της Διεκκλησιαστικής Επιτροπής Ειρήνης και Δικαιοσύνης ε, που θα μας παρουσιάσει την ε, υπόθεση της Κολομβίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να μοιραστώ εδώ μαζί σας την εμπειρία μας μαζί με τις αυτόχθονες φυλές ε, της Κολομβίας που ε, διεκδικούν αξιοπρεπή ζωή στις δικές τους επικράτειες, στο μέσο ένοπλης σύραξης, ε, στρατιωτικών και παραστρατιωτικών, που πολλές φορές μας έχουν απειλήσει, μας έχουν εκτοπίσει, δολοφονήσει, εξαφανίσει, μας έχουν καταχραστεί σεξουαλικά με τη συνενοχή των κρατικών θεσμών για να μπορέσουν να αρπάξουν τη γη μας και τα δικαιώματα μας. Είναι πολύ ιδία η υπόθεση της γης. Στις 16, 8 Αυγούστου του 2012 οι παραστατιωτικοί του ε, ΜΕΤΑ έβαλαν ε, σε ένα στο στόχο ε, τους αδερφούς μας από δύο φυλές και τους έβαλαν ε, μαζί με τους εκπροσώπους της επιχείρησης ε, οι ένοπλοι ζήτησαν λοιπόν γιατί υποχώρησαν από αυτή τη γη που τους ανήκε ε, οι παραστατική στους παραστατικούς και προσπάθησαν να ανακτήσουν αυτές τις γης που προέρχονταν από τους ε, πατέρες τους, τους παππούδες τους που τους είχαν απελευθερώσει την δεκαετία του 50 σε μια συμφωνία που είχε γίνει στο 53 15 χρόνια μετά ε, ακόμα ε, μέλη της οικογένειας αυτής, ε, των οικογενειών αυτών δολοφονούνται. Αλλά εκείνες, εκείνα τα μέρη έγιναν γνωστά γιατί δολοφονήθηκαν ολόκληρες οικογένειες για να πάρει τον έλεγχο η Ισπανοϊταλική εταιρεία Πολυγκρό σε εκείνες τις περιοχές. 12.500 κόσμος ε, εκτοπίστηκαν ανάμεσα στο, 2000, ε, ε, στο συγγνώμη, 1997 και το 2007 αυτές ε, οι επιχειρήσεις ε, θέτουν σε κίνδυνο τους λαούς ε, Σιού και, φελιπάν, την ισορροπία των υδάτων στην περιοχή θέτουν σε κίνδυνο διάφορες, διάφορα είδη ζώων και φυτών που είναι υπό απειλή εξαφάνισης. Αν πάμε στην άλλη άκρη της ε, Κολομβίας, ε, στα σύνορα με τον Παναμά και πάλι οι ε, παραστηριωτικοί παρενέβησαν εκεί. Το 2014 σε νομική απόφαση ε, ε, για, καταδικάστηκαν για εκτοπισμό, για σοβαρή επιβάρυνση της περιοχής και στην δικαστική απόφαση λέει ότι το στη λειτουργία της αυτή η παραστατιωτική οργάνωση ε, καθώς και άλλοι οι οποίοι συμμετείχαν σε επιχειρήσεις ε, θέλησαν να εκτοπίσουν ε, τους τοπικούς πληθυσμούς λόγω του μεγάλου οικονομικού δυναμικού αυτής της επικράτειας. Το 2004 καταγγέλθηκαν οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εμφανίστηκαν από το 1996. Δολοφονήθηκαν 142 άνθρωποι, 136 ήταν στρατιωτικοί και παραστατικοί θύνοντες και 7 από τους αντάρτες του ΦΑΡΚΑ. Δεκατε... Ε, η... Η... Ο κόσμος έχει απογοητευτεί από την... τον εκτοπισμό και βλέποντας τη γη τους να είναι στα χέρια των ε, μεγάλων αυτών επιχειρήσεων. Ε, το Συνταγματικό Δικαστήριο της ε, Κολομβίας στην απόφασή του ορίζει την επιστροφή των γιών αυτών στις κοινότητες που τις είχαν πατροπαράδοτα, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί η συγκεκριμένη απόφαση διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρηματίες από εκεί που καλλιεργούσαν, ε, ε, έκαναν καλλιέργειες φινικέλαιου μετατράπηκαν σε ε, μπανανοκαλλιεργητές. Η Μπανακόλ που είναι θηγατρική της Τσικίτα που είναι γνωστή πολυεθνική εταιρεία ε, έχει καταπατήσει όλες τις γέες μετά, λίγο μετά που αναγκαστικά εκτοπίστηκαν οι τοπικοί πληθυσμοί. Το ίδιο και για την Ουνιβάν που εξάγει προς την Ευρώπη υπό το σήμα Ουρμπάν. Υπάρχουν ε, φοβερές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκτοπισμοί και σε περιοχές ε, όπου λειτουργούν εξορυκτικές βιομηχανίες για την άντληση πετρελαίου, για την εξόρυξη χρυσού και άνθρακα. Επίσης, ε, εκεί όπου γίνονται δρόμοι, υδροελεκτικά εργοστάσια, ε, η επιβεβαίωση των δικαιωμάτων των κοινοτήτων ε, στο μέσο του τρόμου αυτές οι κοινότητες άρχισαν να οργανώνονται για να αποκαλύψουν τις βαθύτερες πηγές αυτών των συγκρούσεων. Συγκρούσεις για λόγω των γεών και βρήκαν, οργανώθηκαν, αντιστάθηκαν και δημιουργήσαν τους δικούς τους μηχανισμούς αυτοπροστασίας και έτσι δημιουργήθηκαν ανθρωπιστικές ζώνες, ζώνες καταφύγια, συγκεκριμένες ζώνες ανθρωπιστικές και χώροι ανθρωπιστικοί μηχανισμοί για να προστατευτεί η ζωή ε, σε περίπτωση χρήσης βίας σε στρατιωτικές και παραστρατιωτικές ε, επιχειρήσεις. Επίσης δημιούργησαν ε, ζώνες βιοπικιλότητας, μηχανισμούς για να προστατευτεί το περιβάλλον. Αυτοί οι μηχανισμοί αυτοπροστασίας συγκεκριμενοποιούν το ανθρωπιστικό δίκαιο και είναι έκφραση της δημιουργικότητας και της αυτονομίας των κοινοτήτων ε, επιτόπου ε, συνοδεύουμε και παρακολουθούμε ως μηχανισμός προστασίας εμείς η Διεκκλησιαστική Επιτροπή Δικαιοσύνης και Ειρήνης και μπορέσαμε έτσι να βοηθήσουμε στην δρέωση τέτοιων σχεδίων. Ο ρόλος τώρα της διεθνούς κοινότητας. Ο ρόλος της διεθνούς κοινότητας ήταν πολύτιμος γιατί οι ε, καταπατητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι υποστηρικτές των παραστρατιωτικών οργανώσεων και η συνένοχή τους ε, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διεθνής κοινότητα έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει να συνεχίσει να παίζει τον ίδιο ρόλο. Η πραγματική παρουσία επί τόπου λειτουργεί ω αποτροπή ε, οι επισκέψεις ασπούσεις επίσης ε, βουλευτών, ε, διακρατικών οργανισμών, οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενισχύουν τα θύματα με, τη, με αυτή τους την παρουσία και οι θύτες ε, αισθάνονται ότι τους παρακολουθεί κάποιος και έτσι οι κολομιανές αρχές αναγκάζονται να εφαρμόσουν κάποιες από τις διεθνείς αποφάσεις. Οι ηγέτες κοινωνικοί αλλά και οι ηγέτες για τα περιβαλλοντικά θέματα είναι σημαντικό να μεταβαίνουν στη χώρα τα ανακοινοθέντα, τα ψηφίσματα διαβιβάζονται στις αρχές Επίσης, ε, η ενημέρωση για το τι κάνουν οι επιχειρήσεις οι ευρωπαϊκές, αλλά και αυτές που εξάγουν προϊόντα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρακολουθούν ε, τι συμβαίνει για να ε, υπάρχει εγγύηση πως οι πόροι που στέλνετε φτάνουν στους δικαιούχους και αποφεύγεται η διαφθορά. Η εφαρμογή των ρητρών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπάρχουν στις εμπορικές συμφωνίες που έχει υπογράψει η Κολομβία ανάμεσα στο 2000 2010 και το 2014 υπήρχε ένα πρόγραμμα για την προστασία και την επιστροφή των γεών στην κοινότητα των Κουρμπαραδό, ε, μίας από αυτές που είχαν εκτοπιστεί. Να σας πω δύο λόγια για το τι γίνεται τώρα στην Κολομβία. Προχωράμε προς την πάυση της ένοπλη σύρρεξη με τους αντάρτες της ΦΑΡΚ και φαίνεται ε, να σταματούν τα πλέον η ένοπλη σύρρεξη. Δεν είναι ειρήνη, αλλά είναι ένα απαραίτητο βήμα για να μπορέσει να ενωθεί πάλι μια κοινωνία, να ξεπεράσει την, ε, την ένοπλη βία και να μπορέσει έτσι να ξεπεράσει τις βαθιές κοινωνικές ε, ανισότητες και τη διαφθορά. Για τις αγροτικές κοινωνίες που έμειναν χωρίς γη είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική έγκριση του νόμου Σίδρης για τις σεζόνες της υπαίθρου. γιατί είναι ένα πρώτο βήμα για μια συμφωνία, την υλοποίηση μάλλον της συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους Φάρκα Αναγνωρίζει δικαιώματα αλλά και ε, την ενοχή των όσων συνεργάστηκαν με τους παραστατητικούς. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη στη ε, Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και τη ΦΑΡΚ. Ελπίζω πως το ίδιο θα γίνει και με τις ε, παραστατητικές οργανώσεις. Έχουμε τέλος και απαιτούμε να υπάρξουν μηχανισμοί ελέγχου έτσι ώστε οι εταιρείε οι ευρωπαϊκές ή αυτές που έχουν επαφές με την Ευρώπη να μην μπορούν να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή να είναι συνένοχοι και ωφελούμενοι από αυτές τις παραβιάσεις. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανοηρεύομαι ε, οι άνθρωποι να μάθουμε τα διδάγματα του παρελθόντος και εμείς έχουμε μάθει ότι οι κοινωνικές ε, σειράξεις μπορούν να ξεπαραστούν. δεν είμαστε απογοητευμένοι λόγω της ανθρώπινης βαρβαρότητας ε, και των συνεπειών της τεράστιες και δυνατές ε, παντοδύναμες εταιρείες έχουν καταστρέψει το περιβάλλον μόνο και μόνο για κέρδη και πιστεύουν ότι οι ίδιες δεν θα επηρεαστούν. Για το καλό της ανθρωπότητας μάλιστα έλεγαν ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν την βία κατά των κακών. Η πραγματικότητα όμως αποδυναμώνει το μήνυμά τους. Εάν εμείς αγωνιστούμε για τη δικαιοσύνη, την κοινωνική και την περιβαλλοντική σε όλες τις γωνίες της γης, δεν θα έχουμε μόνο πιο ασφαλή κόσμο, ασφαλή γη, αλλά θα έχουμε ένα ανθρώπινο μέλλον. α ενωθούμε στο δρόμο για μια αξιοπρεπή ζωή για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη. Εσείς οι βουλευτές από εδώ μπορείτε να δώσετε, να κάνετε σημαντικά βήματα και ίσως να ζητήσω με όλο το σεβασμό να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα 28 ανθρώπους που δολοφονήθηκαν βία φέτος μόνο. Πολλοί από αυτού ηγέτε κοινωνικοί, υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβαλλοντικών δικαιωμάτων που δολοφονήθηκαν επειδή ονειρεύτηκαν ένα πιο δίκαιο κόσμο. Για του δολοφονηθέντε ε, ολόκληρο τον κόσμο, επειδή δούλευαν για έναν καλύτερο κόσμο, πιο ανθρώπινο. Για του συντρόφου και συντρόφισε που μπροστά στη δουλειά για τα ανθρώπινα δικαιώματα Εκείνου που συνοδεύονται θύματα στην Κολομβία, ηγέτε κοινωνικού που εργάζονται για ένα πιο δίκαιο κόσμο, για μια χώρα πιο δίκαιη και για τους εργαζόμενους για την ειρήνη. Νομίζω ότι μπροστά στις δολοφονικές σφαίρες είναι σημαντικό να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Muchas gracias. Bueno, Ευχαριστώ. Τέλος θα δώσω το λόγο στον τελευταίο μας προσκεκλημένο για απόψε, τον κύριο Αλή Κάμπα, που θα μας διηγηθεί και θα καταγγείλει τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του, τη Λιβερία. Παρακαλώ κύριε Καμπά και σας αφήνω με την Αντιπρόεδρο ε, Μπεθέρα. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω σήμερα. Αλή Καμπά λέγομαι από τη Λιβερία. Εργάζομαι με το Ίδρυμα Αϊφόρου Ανάπτυξης ε, και συνεργαζόμαστε με κοινότητες της Υπέθρου στην Λιβερία για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους στη γη και στους ε, πόρους. Εγώ εστιάζω στα δικαιώματα της γης Συνεργαζόμαστε όπως είπαμε με τις κοινότητες της Υπέθρου αλλά και με το κράτος για να αναπτύξουμε πολιτικές οι οποίες αναγνωρίζουν τα δικαιώματα αυτά. Η παρουσίασή μου σήμερα θα εστιαστεί σε πέντε σημεία. Πρώτον, να σας πω το να σας παρουσιάσω το πλαίσιο στο οποίο γίνεται η αρπαγή γης, αλλά και οι συναλλαγές στην ε, Λιβερία, εμπειρίες, επιτόπιες από τη δουλειά που κάνουμε. Ε, επίσης, ε, να αναφέρω την εμπλοκή Ευρωπαίων επενδυτών σε τέτοιες συναλλαγές στη Λιβερία και κάποιες από τις προσπάθειες που κάνουμε στη Λιβερία για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές και να κάνω και κάποιες συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πλαίσιο στη Λιβερία δεν διαφέρει πολύ από αυτά τα οποία είπαν εδώ οι συνάδελφοι. Έχουμε ένα σύστημα ασθενές όσον αφορά τα δικαιώματα στη γη. Υπάρχει ένα διπλό, διτό νομικό σύστημα το οποίο δεν σέβεται τα εθνικά δικαιώματα. Η γη βεβαίως ε, κατά κανόνα είναι στην ιδιοκτησία είτε κάποιων που κατοικούν στη πόλεις ή στα χέρια του κράτους και έχουμε ένα πολύ επίση άσχημο ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά την καλλιέργεια γης. Δεν έχουμε κάποια ολοκληρωμένη αγροτική πολιτική ούτε κάποιο θεσμικό όργανο στο οποίο μπορεί κανείς να προσφύγει αν δεν συμφωνεί με κάτι το οποίο γίνεται στην Λιβερία. Τα κέρδη τα οποία προκύπτουν, οι πρόσοδοι μέσω των παραχωρήσεων ε, και των αδειών εκμετάλλευσης ε, διανέμονται με τρόπο ισότιμο ε, οι περισσότεροι από αυτούς που υποφέρουν από άδειες παραχώρησης δεν λαμβάνουν επαρκείς αποζημιώσεις. Τώρα θα ήθελα να σας αναφέρω μια συγκεκριμένη περίπτωση μια εταιρεία που λέγεται Google, Valeria Liberia που ανοίξει μια άλλη εταιρεία που λέγεται Gullin Agro Resources. Όπως είπα, δεν υπάρχει πραγματική προστασία των δικαιωμάτων αυτών και το κράτος έχει δώσει πάνω από 300.000 εκτάρια γης ε, στην εταιρεία αυτή, την ε, GVA. Και σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά στην περιφέρεια Tarjewon, βλέπουμε πως η εταιρεία, η GVL, έχει πρόσβαση στην γη χωρίς να έρθει πρώτα απ' όλα σε συνεννόηση με τις τοπικές αυτές κοινότητες και βεβαίως ε, έχουμε και ξεκάθαρη αρπαγή της ε, γης και στις περιπτώσεις στις οποίες ε, υπήρξε κάποια αντίσταση η εταιρεία χρησιμοποίησε κάποια μέσα με τα οποία εξανάγκασε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που ήθελε μέσω πολιτικής πίεσης, παραδείγματος χάρη. Η εταιρεία ήρθε σε επαφή με τους πολιτικούς στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για να εξαναγκάσει την κοινότητα είτε να φύγει από τη γη, είτε να υπογράψει για την χρήση αυτή, είτε απλά τους ε, διώχνουν από εκεί. Είχαμε περίπτωση στην οποία ένας ε, επόπτης, ε, θα έλεγα, δεν ξέρω τι είναι συγκρίσιμο εδώ πέρα, διοικητής μιας περιφέρειας απείλησε διάφορους ε, προεστού, θα λέγαμε, μια κοινότητα και είπε ότι θα έπρεπε να πείσουν την κοινότητα να συνυπογράψει, αλλιώ θα χάσουν τι δουλειέ του. Οπότε, ακόμα και αν ε, προσπαθούσε κάποιος να αντισταθεί σε αυτές τις ε, εξαναγκαστικές τακτικές υπήρχε και εκφοβισμός. Υπό την έννοια ότι δεν ε, θα είχαν ε, δουλειές κάποια μέλη της ε, κοινότητας. Και αν δεν λειτουργήσει και αυτό, βλέπουμε απειλές σε κάποιες από αυτές τις περιοχές. Έχουμε δει και παραστρατιωτικούς οπλισμένους φύλακες να μπαίνουν στις κοινότητες για να επιβάλλουν να εφαρμόσουν αυτά τα συμβόλαια. Και κάποιοι έχουν πεθάνει και τραυματιστεί. Οπότε περισσότεροι άνθρωποι εκεί πέρα είναι ευάλωτοι σε τέτοιες συναλλαγές. Ο αντίκτυπος αυτός ε, έχει ήδη καταγραφεί και από τους συναδέλφους. Στην περίπτωσή μας οι άνθρωποι εκδιώκονται από την γη, χάσαν την καλλιεργήσιμη γη και δεν μπορούν άρα να επιβιώσουν να βγάλουν τα προς το ζήν. Υπήρχε και βεβήλωση ιερών τόπων και τα γυναικόπαιδα βεβαίως ε, είναι ακόμη πιο ευάλωτα. Υπάρχει το θέμα βεβαίως ε, της αποδάσωσης, ε, της καταστροφής υδροτόπων, της ρήπανσης κατακαιρματισμού των κοινοτήτων και μετά δημιουργούνται συγκρούσεις και φτώχεια. Αυτές είναι κάποιες από τις προκλήσεις που είχαμε στη Λιβερία και τις έχουμε καταγράψει. Τώρα. Οι Λιβεριανοί, ή Μικιό, και τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων προσπάθησαν να αντισταθούν σε αυτά τα πράγματα, αλλά οι επενδύσεις είναι μεγάλες και η επιρροή επίσης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επενδυτές από την Ευρώπη έχουν εδώ πέρα μεγάλο μερίδιο ευθύνη. Πάνω από 25% των ε, κονδυλίων που πηγαίνουν στην ε, GVL ή e GAR, GAR ε, προέρχονται από την Ευρώπη. Και εδώ πέρα βλέπετε κάποιες τράπεζες που έχουν επενδύσει στην GAR. Οι επενδύσεις αυτές τελικά μέσω της GAR επηρεάζουν τις κοινότητες της ε, Λιβερίας. Όπως είπα λοιπόν, στην ε, Λιβερία υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, απαιτούν τα δικαιώματά τους οι κοινότητες, αλλά υπάρχει ένα νομικό κενό και πολιτική πίεση ταυτόχρονα και όπως είπα είναι και κατακαιρματισμένες οι κοινότητες, οπότε παρά τις προσπάθειες εξακολουθούν να χάνουν τα δικαιώματά τους. Έχουμε τοπικές ΜΚΟ, έχουμε συνεργαστεί με το κράτος να αναπτύξουμε πολιτικές, έχουμε χρησιμοποιήσει διεθνή μέσα αλλά τα αποτελέσματα είναι πάντα πένιχρά γιατί εξακολουθούν να χάνουν την γη τους οι κοινότητες. Συνεργαζόμαστε με διεθνείς εταίρους, με οργανώσεις όπως το Friends of the Earth, Global Witness, για να ασκήσουν πίεση σε κάποιους από τους χρηματοδότες και βλέπουμε πως παρόλες τις προσπάθειες αυτές οι εταιρείες δεν εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, δεν χρησιμοποιούν τα διεθνή μέσα για να σεβαστούν τα εθνικά δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και πάλι στα ίδια καταλήγουμε. Αυτές είναι οι προκλήσεις και έχουμε τις εξής συστάσεις να κάνουμε. Είναι απλές, αλλά πολύ σημαντικές για τις ε, τοπικές κοινότητες στη Λιβερία και ίσως αλλού στην Αφρική. Θεωρούμε πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενισχύσει τους ε, δεσμευτικούς κανονισμούς για τις ευρωπαϊκές εταιρείε οι οποίες επενδύουν στις κοινότητές μας. Θεωρούμε επίσης πως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, επιβάλλει κάποιους κανονισμούς ε, και να υιοθετήσει διάφορα μέσα του ΟΗΕ για να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν λειτουργούν στις ε, κοινότητές μας διάφορες εταιρείε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και τους διοργανωτές για την ευκαιρία που μου έδωσαν να μιλήσω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους ε, τους ομιλητές. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο άμεσα στους συναδέλφους γιατί έχουμε λίγη καθυστέρηση και δεν θα ήθελα ε, να μείνει κανείς εκτός, να μην προλάβει να παρέμβει. Ξεκινάμε λοιπόν με τον ε, κύριο Ντεμεσμάκερ. Κύριε Ντεμεσμάκερ, Παρακαλώ να είστε σύντομοι. γιατί έχουμε και παρεμβάσεις της εξωτερικής υπηρεσίας και τα λοιπά και τα λοιπά, οπότε ένα λεπτό περίπου, κάντε ό,τι μπορείτε. Θα προσπαθήσω στα Ολλανδικά βεβαίω. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ και ειδικά τους προσκεκλημένους μας από τη Λατινική Αμερική και την Αφρική. Οι εμπειρίες και οι μαρτυρίες, οι επιτόπιες βεβαίως είναι πάρα πολύ δυνατές. Σας ευχαριστώ και καλώς ήρθατε στις Βρυξέλλες. Κυρία Κασέρες, όλοι συγκλονιστήκαμε από τον θάνατο της μητέρας σας, του Νέλσον Γκαρσίας και πολλών άλλων και θεωρώ πως μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε με την έκκληση στις αρχές της Ονδούρας να κάνουν κάτι να κινητοποιηθούν για να τελειώσει η ατιμορρησία. το δικαίωμα στην καλλιεργήσιμη γη οπωσδήποτε για τους αγρότες της αναπτυσσόμενες χώρες είναι ο πυρήνας της οι τους. Ε, εκεί πέρα βγάζουν τρόφιμα για να ζήσουν και να πουλήσουν ε, στην τοπική αγορά και βεβαίως ε, συχνά βλέπουμε πως εκδιώκονται δια της βίας από την γη τους και η Oxfam και απευθύνομαι τώρα προς την κυρία Σάρινεν ήταν μια κινητήριος δύναμη για την κύρωση της εθελοντικής οδηγίας για την διαχείριση δασών και γεών από την Επιτροπή Διατροφικής Ασφάλειας του ΕΦΙΟΥ του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ το ερώτημα είναι κατά πόσον εφαρμόζεται βεβαίως και πώς μπορεί να βελτιωθεί η εφαρμογή του κανονισμού αυτού γνωρίζοντας πως ε, τα κράτη-μέλη, παραδείγματο χάρη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και η Παγκόσμια Τράπεζα, κατά πόσον τα μεταφράζουν αυτά στην πράξη σε καλύτερη πολιτική. Επίσης, ε, τον Οκτώβριο του 2012 ξεκίνησε η Oxfam μια σχετική καμπάνια για να σταματήσει η αρπαγή γης στις αναψώμενες χώρες. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει αντιδράσει μέχρι σήμερα και αν ναι με ποιον τρόπο. Βλέπω ο χρόνος πιέζει, έχω και άλλες ερωτήσεις, θα περιμένω τον επόμενο γύρο. Ευχαριστώ, πολύ κύριε Δημασμανικέρε. Η κυρία Ουρρίκη Λούνατσικ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ επίσης για τις μαρτυρίες όλων όσων μιλήσατε και εγώ θέλω μαζί σας να εκφράσω τη λύπη μου για την δολοφονία της Μπέρτα Κάσερες αλλά και όλων των υπολείπων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ονδούρα, στην Κολομβία, στη Λιβερία και σε όλα τα άλλα μέρη του κόσμου. Εγώ ε, μετέβη το 2013 με την ειδική αποστολή του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να παρακολουθήσουμε τις εκλογές τότε. Γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση εκεί. Για να είμαι σύντομη, έχω να κάνω δύο ερωτήσεις ε, κατά βάση. Η μία, ε, την μία απευθύνω στην εκπρόσωπο της FMO, της ε, Ολλανδικής Επενδυτικής Τράπεζας, τράπεζα Επενδύσεων, γιατί μας καλέσατε να σας υποβάλουμε προτάσεις για βελτίωση της συμπεριφοράς σας. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο έχουμε ζητήσει από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι η δημιουργία ενός είδους καταπιστεύματος, trust fund, ε, των επενδυτικών ε, θεσμών για να υποστηρίζονται οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι αυτό κάτι το οποίο έχετε φανταστεί ότι μπορεί να φτιαχτεί μαζί με άλλες ε, επενδυτικές εταιρείες οι τράπεζε που επενδύουν στι διάφορε χώρε ώστε να υποστηρίζονται οι υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω πως αυτό ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Πέρα από τα όσα είπατε εσεί, ότι δηλαδή Ο επενδυτή είναι έτοιμο όχι μόνο να διαπραγματευτεί, αλλά να στηρίξει και τους υποστηριχτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δεύτερο στοιχείο είναι Ίσως ε, καλύτερα να απευθύνω αυτήν την ερώτηση στον πρέσβη της Ονδούρας που είναι εδώ και από τον οποίο γνωρίζω. Κάτι το οποίο ζητήσαμε με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της περασμένης εβδομάδας είναι με την ε, Αμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία συνεργαζόμαστε, αυτό που ζητήσαμε και αυτό που πραγματικά πιστεύω ότι θα ήταν εξαιρετικό να γίνει είναι ένα είδος έρευνας, ανεξάρτητης έρευνας, όπως ε, γίνεται στο Μεξικό με την Αμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όχι μόνο με κάποιους ανθρώπους, αλλά μια ανεξάρτητη έρευνα που θα προσπαθήσει όντως να διευκρινίσει πριν ήταν οι δράστες της δολοφονίας της Μπέρτα Κάσερες και όλων των υπολείπων. Και επίσης ε, μέχρι την ε, ηγεσία, όλη την, την κλίκα. Για να το πούμε έτσι, και, γιατί εδώ η Μπέρτα Θουνίκα μας είπε ότι η Μπέρτα Κασέρες είχε επιληθεί δημόσια 33 φορές και ότι όλες αυτές οι επιλέσεις ήταν συνδεδεμένες με την κατάσταση. Και η Ρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω στα γερμανικά και ευχαριστώ όλους τους συζητητές ε, για την ενδιαφέρουσα ανάλυση ε, που μας δώσανε αλλά και τις συμβουλές τους. Ακούσαμε για παράδειγμα ότι η Λατινική Αμερική και η Αφρική ε, κάνουν δουλειά που αφορά και την αποστολή για την Ασία όπως είναι για παράδειγμα η Μιανμάρ και η Καμπότζη είναι ένα παγκόσμιο λοιπόν φαινόμενο ε, και τα όλα ασκούσαμε λοιπόν. Θα ήθελα να γύρω το ε, ερώτημα για ποιο λόγο στο σχέδιο δράσης ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα το ζήτημα κατοχής γης δεν αναφέρεται επαρκώς. Έχουμε ένα πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αγωνίζονται για τα δικαιώματα κατοχής γης και εσείς μας αναφέρατε τις ε, διάφορες, ε, ε, τους διάφορους παράγοντες και τους κινδύνους. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να επιχρεώσουμε εκτενέστερα. Θέλω να ρωτήσω κάτι και στον πρέσβη από, τον, από, τη Χονδού, από τη Χονδούρα. Η συνάδελφός μου το ανέφερε και είδα ότι η κυρία Κασέρος το ζητήσατε και εσείς να υπάρξει μια ανεξάρτητη έρευνα αυτή, αυτών των δολοφονιών από την ε, πρεσβεία μας ε, δώσατε έγγραφο όπου λέτε τι ακριβώς έχετε κάνει, όμως διαβάζοντάς το αναρωτιέμαι ότι εσείς μιλήσατε ε, με τον Γενικό Διευθυντή των Αμερικανικών, κρατών και θα χρησιμοποιηθούν τα μέσα της Επιτροπής κατά της Διευθοράς. Εγώ διαβάζοντάς το όμως δεν βλέπω ότι ασχολείται με φόνους αλλά με τη Διευθορά και πιστεύω λοιπόν ότι είναι είναι σημαντικό η Αμερικανική Επιτροπή να κάνει μια έρευνα για αυτές τις δολοφονίες και να μην δημιουργηθεί κάτι διαφορετικό το οποίο συνδέεται με την Επιτροπή η οποία έχει εντελώ διαφορετική εντολή. Ίσως λοιπόν ο κύριος Πρέσβης θα μπορούσε να απαντήσει και πάνω σε αυτό ε, το θέμα. Είναι σημαντικό λοιπόν να επιληθεί το ζήτημα από μια ανεξάρτητη επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λόχπια, ο κύριος Παντσέρη. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι τα όσα ακούσαμε επιβεβαιώνουν ε, την ε, δύσκολη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτές οι μαρτυρίες ε, θα έπρεπε μάλλον να ακουστούν ε, από πολλούς ευρωβουλευτές γιατί έτσι θα συνειδητοποιούσαν πόσο επίγον είναι να γυρίσουμε σελίδα και στις ευρωπαϊκές πολιτικές ξεπερνάντας κάποιες υποκριτικές θέσεις που χαρακτηρίζουν τις ενεργειές μας και αναφέρομαι στο εξή. Καταρχάς θα πρέπει νομίζω να ξαναδούμε και σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν σήμερα εδώ να ξαναεξετάσουμε τη δική Είμαστε μας θέση απέναντι στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και ε, να ε, τονίσουμε του όρου σε αυτέ τι συμφωνίε που συνδέονται με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί πολύ συχνά οι θελημένα αυτέ οι συμφωνίε αφήνουν ε, ε, στο βάθο και στην άκρη τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και έτσι αυτά μετατρέπονται σε πολύ σημαντικό θέμα. Έπειτα νομίζω ότι θα πρέπει να μελετήσουμε κατά κάποιο τρόπο και με τη ευκαιρία των Panama Papers ένα είδο κανονισμού που θα μπορούσαμε να προτείνουμε στη προσυζήτηση για τον ε, υπερβολικό εξοεδαφικό χαρακτήρα των πολυεθνικών εταιριών. Διότι εδώ στην ουσία ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι στην ουσία δεν τηρούνται κανόνες. Και εδώ δεν μιλώ μόνο για την αρπαγή γης, αλλά γενικότερα για τα θέματα των ε, δικαιωμάτων. Είναι δύο τομείς ε, επί των οποίων πρέπει να δράσουμε και να σημειώσουμε αστροφή στις ευρωπαϊκές πολιτικές, γιατί αυτό μας ζητούν οι μάρτυρες που είναι σήμερα εδώ. Τους ευχαριστώ με την ευκαιρία και μάλιστα πρόκειται για πράγματα που συμβαίνουν σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Ευχαριστούμε κύριε Πανζέρη. Τελευταίος ο κύριος Ορμπάν. Και εγώ θα αναφερθώ στην υπόθεση της Ονδούρα και στην υπόθεση της ε, δολοφονίας της Μπέρτα Κάθερες. Ε, ε, καταρχάς, τη συλληπιτήριά μου όχι μόνο για την οικογένειά σας, αλλά και για την Κοπίν. Εγώ ήμουν τμήμα μιας διεθνούς αποστολής μετά από αίτημα της οικογένειας της Μπέρτα και της οργάνωσης Σκοπίν. Είναι αλήθεια πως η κατάσταση από την αρχή, το παραξικόπημα δηλαδή του 2009, επηρεάστηκαν οι πολιτικές εξελέξεις ε, με ιδιαίτερα ε, ανησυχητικό τρόπο, αλλά θα ήθελα να κάνω και μια σειρά ερωτήσεων ε, για να μπορέσω να για να μπορέσει να απαντήσει άμεσα η Μπέρτα. Όσον αφορά τις εμπορικέ συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, πιστεύω ότι αν και είναι ε, ε, ήδη συμπεφωνημένη και, ε, και εφαρμόζεται αυτή η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, πώς επηρεάζεται και πώς γίνεται τέτοια project τα οποία είναι άμεσα κατά της ασφάλειας των υπερσπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αναφέρατε εκεί. Πώς γίνεται να συνεχίζονται, έπειτα ποιοι είναι οι δεσμευτικοί μηχανισμοί που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν έτσι ώστε οι πολυεθνικές εταιρείε να μην μπορούν να λειτουργούν ατιμωρητοί στις διάφορες χώρες. Υπάρχει κάποια επιτροπή ε, μετά από αίτημα του Εκουαδόρα, του ΝΟΙΕ, που εργάζεται πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν αναφέρεσασταν σε αυτό ή αν έχετε κάποια άλλη ευρύτερη ιδέα για το πώς μπορούμε κάτι να κάνουμε. Τέλος, δύο τελευταίες ερωτήσεις πολύ σύντομες. Όσο ήμουν στην, στην Ονδούρα, υπήρξε μια έκκληση από πλευρά των, ανθρω... των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να ερευνήσουμε τα project της συνεργασίας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ονδούρα, όπως το project Ευρωζουστήσια, Ευρωδικαιοσύνη, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να κατασταλούν ε, τέτοιες οργα... κοινωνικές οργανώσεις όπως η ΚΟΠΗΝ. Χρησιμοποιούνται δηλαδή στρεβλά αυτά τα προγράμματα συνεργασίας. Και έπειτα τι μπορεί να κάνει, νομίζετε, ένα τέτοιο κοινοβούλιο όπως το Ευρωκοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ώστε να καταφέρουμε με αποτελεσματικό τρόπο να προστατεύσουμε τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σε χώρες όπως η Κολομβία, η Ονδούρα ή η Λιβερία παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα απλά και μόνο για να υπερασπιστούν ένα αξιοπρεπές μέλλον για τους λαούς τους και για τη γη τους. Ευχαριστώ πολύ. Μου ζητά το λόγο και ο κύριος Γκζίμπ. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Ένα ερώτημα το οποίο θέλω να γύρω έχει τεθεί ήδη, όμως θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν πέρασε ένα ψήφισμα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ονδούρα. Αφορούσε ιδιαίτερο στους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Ποια είναι η δική σας αξιολόγηση λοιπόν να, το θέμα είναι να συγκρίνουμε την κατάσταση στην Ονδούρα με άλλες λατινοαμερικανικές χώρες. Ποια λοιπόν είναι η κατάσταση για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς μπορούν να ε, δουλέψουν σε συνάρτηση ε, με αυτό το οποίο συζητούμε ε, σήμερα, δηλαδή την αρπαγή γης. Είναι ένα φαινόμενο που είναι ιδιαίτερα γνωστό σε αυτό το κοινοβούλιο. Ήδη από την προηγούμενη θητεία, του, θητεία το είχαμε συζητήσει αυτό, το είχαμε συζητήσει στην ε, ετήσια αξιολόγηση για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον πλανήτη. Αυτό λοιπόν επανειλημμένος είναι ένα θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε. Ε, και πάντοτε αντιμετωπίζουμε ε, φαινόμενα όπου κάποια ζητήματα τα συζητούμε εντόνως ε, και όπου περνάμε μια σημαντική φάση και ίσως να έχει φτάσει αυτή η στιγμή και για την αρπαγή γης. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνουμε μια σύγκριση. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω μόνο να κάνω μια σύντομη ερώτηση σε σχέση με τα όσα είπαν οι υπόλοιποι ε, ευρωβουλευτές ε, για όλους τους ομιλητές αλλά και προς την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ποια πιστεύετε ότι είναι, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος ε, του Συμβουλίου και όσον αφορά την όθηση προς τις εταιρείες που εγκαθίστανται στις διάφορες εταιρείες μέσω των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πρεσβειών μας στις χώρες αυτές πώς και αν ε, προωθούν ενεργοά όλα τα στάνταρ που υπάρχουν όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν υπογραφεί εδώ και πέντε χρόνια και που είναι τελικά τελείως εθελοντικά ε, εφαρμόσιμες. Αυτό για το οποίο μιλάμε είναι το απόλυτο παράδειγμα για το πώς η δέσμευση των εταιριών για αυτός ο τρόμος που έχουμε εμείς να, να ζητήσουμε να είναι δεσμευτικά όλα αυτά για τις επιχειρήσεις, τελικά για τις καλές επιχειρήσεις ε, εντάξει, είναι τέλειο. Είναι κάτι που υποτίθεται ότι είναι δεσμευτικό, Υπάρχουν αυτές που ακολουθούν τις καλές πρακτικές, αλλά εκείνες ε, οι οποίες δεν θέλουν μπορούν και να μην τις ε, τηρούν αυτές τις κατευθύνες γραμμές. Και θα δώσω έτσι το λόγο στην Υπηρεσία Εξωτερική Δράση τον κύριο Ρικάρντο Σέρι, που είναι επικεφαλής του Τμήματος Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολιτικές Συνεργασίες. Αν δεν ξέρω αν εσείς θα μιλήσετε μόνο ή αν θα μιλήσετε ε, συνεταιρικά με άλλον συναδελφό σας. Έχετε τέσσερα λεπτά στη διάθεσή σας. Σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν είμαι τμήματάρχης ακριβώς. Λοιπόν, να σας κάνω μια σύντομη εισαγωγή για τα στοιχεία της ε, πολιτικής, για τα θέματα της αρπαγής γης από την δική μας τη Σκοπιά και μετά θα δώσω τον λόγο σε άλλους συναδέλφους που ίσως έχουν να κάνουν σχόλια που αφορούν ειδικά τις ε, χώρες αυτές και τα συγκεκριμένα γεγονότα. Και θα προσπαθήσω να απαντήσω και στο ερώτημα της κυρίας Λοχμπίλερ και άλλων. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για αυτή την συζήτηση γιατί είναι επίκαιρη και πολύ σημαντική για να δώσουμε σημασία σε αυτό το ζήτημα. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν Υπήρχε μια έκθεση που δημοσιεύτηκε πέρσι για την αρπαγή γης που μας ενέπνευσε όσον αφορά το σχέδιο δράσης για ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία. Υπάρχει ένα έγγραφο πολιτικής ε, το οποίο καλύπτει διάφορα ζητήματα Και νομίζω πως ε, επίσης βεβαίως απαντάμε έτσι και στο ερώτημα της κυρίας ε, Λοχμπίλερ. Ίσως όχι επαρκώς, αλλά σύμφωνα με την ε, δική σας την ερμηνεία, αλλά οπωσδήποτε πολύ πιο συγκεκριμένα από ό,τι παρελθόν. Και μάλιστα γίνεται και από διαφορετικές σκοπιές από τη σκοπιά των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ξέρετε τι σημασία αποδίδουμε σε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Κομισιόν και βεβαίως με το να εστιάζουμε ειδικά στην αρπαγή γης και στα λοιπά δικαιώματα της γης ε, των αυτοχθόνων ε, είναι κάτι το οποίο βεβαίως έχει μεγάλη σημασία και με αυτό σχετίζεται και το σχέδιο δράση για τους ίδιους τους αυτόχθονες λαούς και οι δράσεις που αναπτύσσονται. Θα υπάρξει ένα νέο έγγραφο που συντάσσουμε αυτή τη στιγμή για να ξανα ξεκινήσουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Αυτόχρονους λαούς, ειδικά όσον αφορά την ε, ελεύθερη πρώτερη συνένεση που αναφέρθηκε για να εφαρμόζεται όπως υπόθηκε. Άλλα ζητήματα που θα ήθελα να αναφέρω σύντομα είναι βεβαίως το ενδιαφέρον και η στήριξή μας για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευρά επιχειρήσεων και κάποιων κατευθυντηρίων αρχών. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που σχετίζονται με αυτό. Όπως ξέρετε τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν εθνικά σχέδια δράσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα δημιουργήσει μια νέα πολιτική και δίνουμε βάση στο πιο κρίσιμο ζήτημα κατά την απόψή μας το οποίο είναι η δυνατότητα προσφυγής που δεν είναι κάτι το δεδομένο αυτή τη στιγμή και η Ολλανδική Προεδρία είναι ιδιαίτερο ενεργή το εξάμεινο αυτό για τα συμπεράσματα και για την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον συναδελφό μου γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ναι, εσεί ολοκληρώσατε, καταναλώσατε το χρόνο που σα είχα δώσει, αλλά παρακαλώ πάρτε και εσεί το λόγο για να μα δώσετε μια εικόνα ω επικεφαλή του τμήματο για την ε, Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Έχουμε παρακολουθήσει στενά την κατάσταση στην Ονδούρα και έχουν ε, γίνει αρκετές ε, ε, δηλώσεις πάνω σε αυτό το θέμα, ιδιαίτερω για να κατεδικάσουμε τι απειλέ δολοφονίες και πράξεις βίας. Για παράδειγμα έχουμε την διακήρυξη στην περίπτωση της δολοφονίας της Μπέρθα Κάσερες και του Γκαρσία δεν είναι μονάχα μια ε, διακήρυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερο ε, εταίρο ε, στην Ονδούρα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν τα προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το PDH για παράδειγμα, το οποίο έχει λάβει 5,5 εκατομμύρια ε, και ε, βοηθά στη σύνταξη του εθνικού, ε, του, της Εθνικής Νομοθεσίας για την Προστασία Δημοσιογράφων και έχουμε το έργο Ζουστίσια, το οποίο κόστησε 51 εκατομμύριο ευρώ και θέλουμε να καταλάβουμε πώς ένα έργο το οποίο έχει ως στόχο να υποστηρίξει το νομικό σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ότι χρησιμοποιείται για να καταπιέσει ε, οργανισμούς ε, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά τις Ονδούρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε 40 εκατομμύρια ευρώ από την περίοδο ε, 40 εκατομμύρια για να υποστηρίξει το κράτος δικαίου και την νομοθεσία στη χώρα. Επίσης υπάρχει μια άμεση ε, προστασία ε, προς τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε μια ομάδα η οποία συνεργάζεται με τις πρεσβείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ονόματι Γκρούπο Ενλάσε και έχει έναν διάλογο με τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναλαμβάνει υποθέσεις προς την κυβέρνηση το πρώτο άτομο λοιπόν με το οποίο συναντήθηκε η, κυρία, ε, η ομάδα αυτή ήταν η κυρία Χερμάτα. Αναλάβαμε λοιπόν την ευθύνη ε, ώστε η Αμερικανική ε, Οργανώση να ξεκινήσει μία έρευνα μια ανεξάρτητη έρευνα απέναντι σε αυτήν την υπόθεση και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποστηρίξει μια τέτοια έρευνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίες. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ρινάλντι και τον κύριο Κίνος. Ποιος θα παρέμβει και οι δύο. Μπορείτε να πάρετε το λόγο και οι δύο αν το επιθυμείτε. Η κυρία Ρινάλντι είναι επικεφαλής του τμήματος ε, για τη διακυβέρνηση, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε και τον διευθυντή του τμήματος για την ανάπτυξη της υπαίθρου και την ε, ε, διατροφή. Μπορείτε να μοιραστείτε μεταξύ σας πέντε λεπτά για αυτό το χρόνο σας δίνω και στους δυο μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη και θα ξεκινήσω παρουσιάζοντας ε, το έργο μας από την πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αρχικά εργαζόμαστε ε, για να, για να βοηθήσουμε τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον ε, πλανήτη και για εμάς λοιπόν είναι γνωστό ένα γνωστό και σημαντικό εργαλείο ώστε ε, να καλύψουμε τα κενά σχετικά με το τι συμβαίνει στα ανθρώπινα δικαιώματα και υπάρχουν αυξανόμενες απειλές απέναντι σε αυτούς τους ε, υπερασπιστές αλλά και φαινόμενα αρπαγής ε, γης από ηθαγενείς πολίτες, από αυτόχθονες Ε, για παράδειγμα, εμείς υποστηρίξαμε την Πέρτα ε, Κασέρ το 2014, αλλά και τους συναδέλφους τους. Χρηματοδοτήσαμε νομική βοήθεια και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να βοηθάμε τη δουλειά της ε, στο Κοπίν, αλλά και, με άλλους, αλλά και άλλους συναδέλφους της. Δεν πρόκειται να αναφερθώ σε όλες τις υποθέσεις τις οποίες, ε, στις οποίες βοηθάμε, γιατί είναι τόσες πολλές, ε, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να τονίσω ότι ασχολούμαστε καθημερινά με τέτοιες υποθέσεις σε όλο τον πλανήτη. Τώρα, ε, πέρα από τις λεπτομέρειες, εμείς βοηθούμε όλο και περισσότερο ζητήματα οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, βοηθούμε ε, οργανώσεις ε, στοχεύοντας να βοηθήσουμε την κοινωνία των πολιτών ε, αλλά και την εφαρμογή της 27ης ε, σύμβασης και φέτος έχουμε το Global Goal που θα ξεκινήσει φέτος το οποίο θα συνεργαστεί επίσης με την κοινωνία των πολιτών με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα επίσης ε, να τονίσω ότι πέρα από τα προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα αρχίζουμε να ενσωματώνουμε ε, την προσέγγιση race-based σε όλα μας τα προγράμματα. Θα χρειαστεί χρόνος, ε, το κάνουμε βήμα-βήμα. Στόχος μας όμως είναι στο τέλος να ε, αφορά το ζήτημα όλα τα επενδυτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την προστασία του, προβ... περιβάλλοντας, τη διατροφική ασφάλεια και φυσικά υποδομές και επενδυτικά προγράμματα. Στόχος αυτής της προσέγγισης ε, για την ανάπτυξη δεν είναι μονάχα να μην ε, βλάψουμε αποτρέποντας ε, τις αρνητικές συνέπειες ε, των αναπτυξιακών προγραμμάτων για τις ντόπιες κοινωνίες, αλλά να κάνουμε το μέγιστο καλό συνεισφέροντας στην πραγματοποίηση, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τοπικές κοινότητες, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο, αλλά και είναι και ο βασικός μας στόχος. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Ονομάζομαι Joachim Κλότ. Η ανάπτυξη είναι το ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Θα ήθελα τώρα ε, να ε, συμφωνήσω με κάποιους ε, συναδέλφους από εδώ. Υπάρχει ελλειπής σεβασμός ε, για τα δικαιώματα και υπάρχει έλλειψη διαφάνειας ε, όσον αφορά ε, τις ανταλλαγές και το εμπόριο γεών και αυτό έχει αρνητικές συνέπειες για τις επενδύσεις. Αυτό ακριβώς είναι στο οποίο στοχεύει η Κομισιόν μαζί με άλλους επενδυτές. Αυτό το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε λοιπόν είναι η έγκριση των ε, κατευθυντηρίων της ε, Γενέβης ε, από το Παγκόσμιο Επιστήμιστικό Πρόγραμμα το 2011. Οι κατευθυντήριες αυτές προβλέπουν πώς να βελτιώσουμε την διακυβέρνηση ε, σχετικά με τα ζητήματα ε, γεών, δασών ε, και αλίας. Επενδύσαμε 60 εκατομμύρια για να προωθήσουμε τις συγκεκριμένες κατευθυντήριες. Μέχρι στιγμής έχουμε προγράμματα τα οποία δραστηριοποιούνται σε 18 αναπτυσσόμενες χώρες, οι περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονται στην Αφρική και είναι η Ήπειρος όπου η αρπαγή ε, γης έχει τη μεγαλύτερη σημασία με βάση τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας. Εργαζόμαστε με αυτά τα προγράμματα σε διάφορα επίπεδα. Ένα πολύ σημαντικό επίπεδο είναι η υποστήριξη των κυβερνήσεων για να βελτιώσουν το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με το ε, ε, με την προστασία αλλά και πώς να εφαρμόσουν την νομοθεσία αυτή. Ταυτόχρονα θέλουμε να υποστηρίξουμε τους ντόπιου παράγοντες ούτω ώστε να ε, συμμετάσχουν ε, στον διάλογο αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμπεριλάβουμε και από τις δύο πλευρές, τόσο από το κυβερνητικό επίπεδο όσο και από την πλευρά ε, των, του ντόπιου πληθυσμού, αυτοί οι οποίοι εποφελούνται ζώντας σε αυτές τις περιοχές. Συνεισφέραμε επίσης στην προετοιμασία των αρχών για την υπεύθυνη επένδυση στη γεωργία. Αυτά λοιπόν υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή ε, για την ε, Ευαισθητιστική Ασφάλεια. Οι αρχές αυτές βασίστηκαν στις ε, ε, εθελοντικές κατευθυντήριες ε, για την υπεύθυνη διαχείριση της κατοχής γης και είναι σημαντικές για αυτούς οι οποίοι κάνουν τις επενδύσεις αλλά και για τους ντόπιους πληθυσμούς. Πέραν τούτου, η ομάδα δωρητών σχετικά με τις γης προετοίμασε το αναλυτικό πλαίσιο για επενδύσεις ε, στην Αφρικανική Γεωργία και αυτό ζητήθηκε συγκεκριμένα από το Συμβούλιο του ΕΕ για την Επιστημιστική Ασφάλεια και με τα χαρά το παρουσιάσαμε πέρσι το καλοκαίρι στην Επιτροπή. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να κλείσετε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήδη έχετε καταναλώσει το χρόνο που σας είχα ε, δώσει. Παρακαλώ, ολοκληρώστε την παρέμβασή σας. Okay, I follow you. Ε, ωραία, θα ακολουθήσω τη συμβουλή σας. Θα έλεγα λοιπόν ότι εργαζόμαστε πάνω σε πολύ ευαίσθητα ε, θέματα, πάνω στην άμυνα, στην ομοθεσία, την ενίσχυση των ντόπιων παραγόντων, ενώ ταυτόχρονα παρέχουμε τις κατευθυντήριες, τις αποστολές μας ώστε να είναι πιο ενεργές ε, και επικοδομητικές στον διάλογο που κάνουν για την αντιμετώπιση αυτών των ε, προβλημάτων με τις κυβερνήσεις των χωρών όπου πηγαίνουν. Ευχαριστώ. Αυτό που θέλω να σας θυμίσω είναι ότι θα θέλαμε να λάβουμε όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε και τις οποίες αναφέρατε και γραπτός, ώστε να μπορέσουμε να τις προωθήσουμε στους βουλευτές και στους συμμετέχοντες σε αυτήν την ακρόαση, έτσι ώστε όλα όσα δεν προλάβατε να πείτε προφορικός να τον τα στείλετε γραπτός. Και τώρα έχουμε την τελευταία φάση όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους πρέσβεις που είναι σήμερα εδώ. Έχουμε τον ε, εξοχότητά του, τον κύριο Μαθήτ, που είναι ο ε, εκπρόσωπο ε, ο πρέσβη μάλλον της Ονδούρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Επίσης τον πρέσβη της Κολομβίας στο Βέλγιο, του Λουξεμβούργο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης μεταξύ μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Εσκίνε, που είναι ο πρέσβης της Γουαταμάλα. Αν έχουμε χρόνο θα σας δώσουμε και σας λίγο το λόγο. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Τσέβα της Ονδούρας για τρία λεπτά παρακαλώ. Πρόεδρε, συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι. Η δολοφονία της Βέρτα Κάσερες είναι ένα έγκλημα κατά όλων ε, των πολιτών της Ονδούρας και κατά των αρχών της ελευθερίας ε, που θεσπίζονται από το Σύνταγμα. Η Βέρτα έχει αποτελέσει ένα σημαντικό κομμάτι της εθνικής μας συνείδησης μέσω του αγώνα της για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ονδούρα, την υπεράσπιση και την προστασία του περιβάλλοντος που είναι επίσης προτεραιότητα της εθνικής μας ατζέντα. Από τότε που συνέβη αυτή η δολοφονία, η κυβέρνηση της Ονδούρας ε, γιατί καταδίκασε, την καταδίκασε κάθετα και έχει ξεκινήσει τη δικασία ώστε να προβεί στι κατάλληλε ενέργειε ώστε να υπάρξει επιστημονική, εξονυχιστική και διαφανή έρευνα έτσι ώστε να συλληφθούν οι δράστε αλλά και οι ηθικοί αυτούργοι. Ε, καθώς και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Το κράτος της Ονδούρας αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου μεμονωμένα ή συλλογικά να προωθήσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πρόθεση αυτών καθώς και των θεμελιωδών ελευθεριών. Τα τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί το νούμερο των δολοφονιών λόγω του οργανωμένου εγκλήματος στην Λατινική Αμερική και στην Ονδούρα. Έχουν υπάρξει πολλές δολοφονίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος, ε, της δικαιοσύνης και άλλων που λόγω του αγώνα τους έχουν έρθει σε σύγκρουση με τα συμφέροντα διαφόρων ε, ομίλων και ομάδων. Δεν θα περάσει ατιμωρητή η δολοφονία της Μπερτακάσερης. Αυτό το φίλουμε στο λαό της Ονδούρας. Η κυβέρνησή μας έχει δεσμευτεί για την επίλυση αυτής της υπόθεσης για να ανακτήσει την εθνική και τη διεθνή εμπιστοσύνη και έτσι ε, πρόκειται για πραγματική ποινική διαδικασία. Όλες οι έρευνες, οι ιατρικές, ιατροδικαστικές, επιστημονικές έχουν ξεκινήσει. Μετά από ε, ε, αίτηση της ε, κυβέρνησης της Ονδούρας κλήθη και εκπρόσωπος του ΟΗΕ και του ΙΣΥΠΑ της Αρμοστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και της και της αποστολής για την καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έφτασε στην Τεγκοπασίλικα αυτή την εβδομάδα. Ε, Είμαστε υπέρ της υπεράσπισης των δικαιωμάτων όλων των ατόμων αλλά και των αυτοχθόνων λαών. Επίσης καλούμε όλες τις οργανώσεις των πολιτών να επαγρυπνούν και να ειδοποιούν για αυτές τις καταστάσεις. Επίσης θα θέλαμε οι ευρωπαϊκές εταιρείες να τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις αυτόχθονες ε, λαούς και όταν θέλουν να εγκατασταθούν στη δική μας ε, επικράτεια. Ε, θέλουμε να προστατεύσουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα και το ε, περιβάλλον. Και μου το επιτρέπετε να απαντήσω στην κυρία Λούνα Σεκ, την αγαπητή μας αντιπρόεδρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει τον, ε, δια, ε, τον, την Αμερικανικό Μηχανισμό Διαφάνειας και κατά της διαφθοράς. Είναι η αποστολή του ΟΗΕΑ. Στις 8 μάλιστα Απριλίου η σύμβουλος του Ιω Κοράλες ε, ήρθε στην ε, Ουάσιγκτον στην Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα να διαπραγματευτεί για ε, βραχυπρόθεσμα ένα μνημόνιο για να βελτιωθεί η εφαρμογή αυτών των μέτρων και δυνατότητες έρευνας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσό. Και τώρα έχετε εσείς το λόγο. Και εσείς για τρία λεπτά. Καταρχά, σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετέχω σε αυτήν την δημόσια ακρόαση για αυτό το τόσο ενδιαφέρον ε, θέμα για την Κολομβία. Ο χρόνο, χρόνος βέβαια είναι πολύ περιορισμένος και φυσικά σας προσκαλώ στην πρεσβεία όποτε θέλετε εσάς και όλους τους ευρωβουλευτές ε, για να συζητήσουμε πιο αναλυτικότερα όλα αυτά τα θέματα. Ε, το 2015 ήταν ε, ε, ο χρόνος όπου είχαμε τις πιο χαμηλό αριθμό ε, δολοφονιών τα τελευταία 30 χρόνια. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ελπίζουμε ότι θα είναι επιτυχής, επιτυχές στο τέλος της διαδικασίας ειρήνευσης. Στο δομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην Κολομβία έχουμε φτιάξει μια επιτροπή υψηλού επίπεδου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στόχο έχει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει πολιτικές σε συνεργασία με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να μπορέσουν ελεύθερα να κάνουν τη δουλειά τους. Ε, υπάρχουν εγγυήσεις όσον αφορά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικαιωμάτων ώστε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην άσκηση του καθήκοντό του. Είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα ανάπτυξης καθώς και δημιουργία του προγράμματος εγγυήσεων ε, καθώς και η ε, η Επιτροπή που δημιουργήθηκε για την προστασία των δικαιωμάτων των ε, γυναικών. Το κράτος και η κοινωνία των πολιτών ε, συσκέφθηκε και συμφωνήσαμε όσον αφορά τις υποθέσεις που πρέπει επιγόντως να διερευνηθούν. Πρόσφατα η εισαγγελία ε, ε, αποφάσισε να φτιάξει μια ειδική ομάδα όσον αφορά τις υποθέσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να ξεπεραστεί η ένοπλη σύραξη αλλά και ε, ο στιγματισμός ε, που ε, υπάρχει μετά από όλα αυτά τα χρόνια ενόπλων σειράξεων. Αυτό όχι μόνο θα ενισχύσει τη δημοκρατία, αλλά θα αποτελέσει και ένα ηθικό θεμέλιο για το νέο μας κράτος, για την κυβέρνηση της Κολομβίας. Τα συμφέροντα, βέβαια, τα εταιρικά είναι πολύ σημαντικά. Το 2014 δημοσιεύθηκε η σύνδεση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις εταιρικέ ευθύνες. Έτσι, ε, μέσα από το διάλογο ε, έχει οικοδομηθεί ε, τα έτη 2012-2013 μία συνεννόηση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι ξένες εταιρείες εκεί. Ε, και όλα αυτά σε συνεργασία με πολυεθνικές, με εταιρείες και με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει να αναφερθώ δε και στην επιστροφή γεών. Είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο η Κολομβία που προχώρησε σε αποζημίωση των θυμάτων και μάλιστα έχει επιστρέψει γεές μετά από τη λήξη της ενόπλης, ε, των, ενόπλ, των ενόπλων σειράξεων. 100.000 εκτάρια πρόκειται να επιστραφούν και γνωρίζουμε Βέβαια ότι είναι πολύ δύσκολο όλα αυτά και θα πρέπει ακόμα να ολοκληρωθούν, αλλά είναι ε, απαραίτητα για να επικρατήσει η ειρήνη στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα κλέψουμε 10 λεπτά από, ε, από το επόμενο θέμα, ώστε οι συμμετέχοντες να δώσουν μια τελευταία απάντηση. Δύο λεπτά έκαστος, αλλά δεν μπορώ παρά να δώσω και ένα λεπτό και το λόγο στον κύριο Σκίνερ. Δεν θέλετε? Ε, εντάξει. Εμείς σας κρατήσαμε πάντως ένα λεπτάκι. Λοιπόν, αρχίσουμε με την αντίστροφη σειρά. Η κυρία Σάρινεν, ναι. ένα με δύο λεπτά για να βγάλετε συμπεράσματα ή να απαντήσετε σε κάποια από τα ερωτήματα που ετέθησαν. Ευχαριστώ πολύ. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο ε, ερώτημα σχετικά με τις κατευθυντήριες. Οι κατευθυντήριες όταν ε, υιοθετήθηκαν το 2012 ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή διότι ήταν ε, πολύ σημαντικές. Αν εφαρμόζονταν τότε όλες οι υποθέσεις αρπαγής γης θα είχαν αποφευχθεί. Ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα το ότι έλαβαν υποστήριξη και αυτή τη στιγμή το ερώτημα είναι πώς θα τις εφαρμόσουμε και αν εφαρμόζονται σε κρατικό επίπεδο και χαίρομαι ιδιαίτερως για τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει ηγετικό ρόλο ώστε να διασφαλίσει πως οι κατευθυντήριες αυτές εφαρμόζονται ιδιαιτέρως όταν επανεξετάζεται η εθνική νομοθεσία σχετικά ε, με τη γη και τους φυσικούς πόρους. έχω παρατηρήσει αρκετά προβλήματα ε, πάνω σε αυτό το θέμα, κυρίως στην Αμερική και γι' αυτό το λόγο περισσότερο πρέπει να γίνουν πάνω σε αυτό. Υπήρξε και ένα ερώτημα σχετικά με την ε, ενασχόληση της Oxfam, τη, σχέση της ε, Oxfam με την Παγκόσμια Τράπεζα όπως και με τη σχέση μας με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουμε ε, ασχολούμαστε με ζητήματα τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων και περιβαλλοντικά ζητήματα. Ε, τα ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πολύ συχνά είναι ανοιχτά στο να υπάρξει διάλογος και παρέχουν ταυτόχρονα συμβουλές με το πώς να αντιμετωπίσουμε τα συγκεκριμένα θέματα. Η αντιπόκριση υπάρχει τώρα πώς θα μεταφραστεί αυτή σε δράση. Εκεί χρειάζεται αρκετή δουλειά. Σας ευχαριστώ. Okay. Σας ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο για τα συμπεράσματά της στην Μπέρτα Θούνιχα Κάσερες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μου ετέθησαν πολλά ερωτήματα, αλλά θα απαντήσω μόνο στα πιο, αυτά που θεωρώ εγώ τα πιο σημαντικά. Το κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό για μας και είναι πολύ δύσκολο να πούμε εμείς τι μπορείτε να κάνετε. Αυτό που θέλουμε είναι να μην ε, ε, να μην ε, ξεχάσετε την κατάσταση που επικρατεί στην Ονδούρα, όπως σας εξηγήσαμε, 48 μέρες ε, έχουν περάσει από τότε που μας αρνήθηκαν επισήμως την συμμετοχή στην έρευνα. Εμείς καταθέσαμε επίσημο αίτημα ενώπιον των αρχών της Ονδούρας που μας αρνούνται την πρόσβαση στις πληροφορίες και έχουμε κάνει και προσφυγή σε αυτήν την απόφαση Ε, είναι μια είναι χώρα όπου δεν εισακουγόμαστε ως θύματα. Δεν παραμελούνται ή αγνοούνται τα αιτήματά μας. Κάνουμε ε, αιτήματα επίσημα όπως μέσω της ΜΑΣΗ που έχει συγκεκριμένη εντολή για τη διαφθορά, κατά της διαφθοράς και όχι ε, για την διερεύνηση κλιμάτων. Η Αμερικανική Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει το δικαίωμα να παρέμβει ε, από πλευρά ε, του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Ερνάντες, έχει λάβει τέτοιο έτοιμο για να ξεκινήσει έρευνα. Σα ευχαριστώ, Μπέρτα. Κυρία Μπροκ Πολύ καλά το προφέρατε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λούνατσεκ έθεσε ένα ερώτημα σχετικά με την FMO. FMO και άλλες αναπτυξιακές τράπεζες και θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό. Είμαστε μια αναπτυξιακή τράπεζα και εντολή μας είναι να επικεντρωθούμε στην, ε, σε έργα του ιδιωτικού τομέα Χρηματοδοτούμε λοιπόν πελάτες οι οποίοι υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη αλλά με έναν κοινωνικό και περιβαλλοντικό τρόπο ταυτόχρονα. Επικεντρώμαστε ε, στην πρόσβαση σε τρόφιμα, ε, θέσεις εργασίας, χρηματοδότηση και έχουμε ε, ασχοληθεί από κοινού άλλους επενδυτές και σε άλλα έργα, έργα όπως είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η ανάπτυξη, τα οποία μπορούν να φέρουν πρόοδο στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε παρατηρούμε ταυτόχρονα ότι δεν επαρκεί πολλές φορές να επικεντρωνόμαστε στα θέματα ε, στα οποία ασχολούνται οι πελάτες μας, αλλά γι' αυτό θέλουμε μια πολυμερή προσέγγιση και γι' αυτό το λόγο απαιτείται συνεργασία και με άλλους παράγοντες όπως είναι για παράδειγμα ΜΚΙΟ, οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ούτως ώστε να επιτευχθεί πρόοδος ε, σε πολύπλοκες καταστάσεις και γι' αυτό το λόγο διακρίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη να ασχοληθούμε ε, πάνω σε αυτό και γι' αυτό το λόγο ευχαριστούμε ε, που υπήρξε η δυνατότητα να έρθουμε εδώ να συζητήσουμε αυτό, να συζητήσουμε ε, και με την κυρία Κασέρες διότι θεωρούμε ότι όταν είμαστε παρόντες, όταν βρισκόμαστε εκεί με τον πελάτη, τότε μπορεί να υπάρξει η ευκαιρία να βρεθεί ένας τρόπος και νιώθουμε υπεύθυνοι στην εξέβρεση λύσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Πατέρα Αλβέρτο Φράγκο, έχετε και εσείς ε, δύο λεπτά για να ε, κλείσετε. Είναι βέβαιο ότι η Κολομβία ζει ε, αυτή τη στιγμή την μείωση της ένοπλης ε, σύραξης. Ε, έχουμε φτάσει ιστορικά νούμερα. Ωστόσο, πρόσφατες έκθεση του ΕΕ δείχνουν ότι 885 επιθέσεις έχουν γίνει κατά 885 υπερασπιστών συμπεριλαμβανομένων 35 γυναικών. Αυτό το λέει ο ΙΕ. Τα νούμερα ξεπερνούν το μέσο όρο δολοφονιών των τελευταίων 15 ετών. Άρα λοιπόν για στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν τα πάμε καθόλου καλά και αυτό έχει, να, έχει σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αρπαγή γης. Εκτιμούμε την ανησυχία σας για τη δημιουργία ενός μηχανισμού προστασίας και για την ε, ε, συγγραφή διεθνούς νομοθεσίας. Οι όμιλοι χρησιμοποιούν μια ατέλειωτη αλυσίδα υποδιαιρέσεων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να καταγραφούν και να αναλάβουν τις ευθύνες οι μητρικές εταιρείε. Είναι δύσκολο να βρούμε νου είναι τριγατική πια. Αυτό λοιπόν πρέπει να μελετηθεί. Να μελετηθεί πώς θα μπορέσουμε να νομοθετήσουμε διεθνώς ώστε να αποφύγουμε ζημιές ε, που δεν θα μπορούν μετά να διορθωθούν. Κάθε φορά δε, που έχουν ε, ε, καταγγελθεί εταιρείε έχουμε διώξεις, ε, δυσφήμιση απειλές και δολοφονίες και είναι πάρα πολύ πολύτιμη η υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και των βουλευτών που στηρίζουν τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους εργαζόμενους υπέρ της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ και για να κλείσω, κλείσουμε θα δώσω το λόγο στον κύριο Καμπά. Έχετε κι εσείς 1,5 λεπτό για να κλείσετε. Και πάλι ευχαριστώ Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Για εμάς στη Λιβερία και στην Αφρική που είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτού του σοβαρού προβλήματος όπως είπαν και οι συνάδελφοι είναι ατυχές το ότι έπρεπε να ταξιδέψουμε τόσο μακριά για να ακουστούν οι φωνές μας επίσης θεωρούμε πως σε αυτό το κτίριο. Ίσως κάποια προβλήματα από τα προβλήματά μας ε, μπορεί να λυθούν. Στην περίπτωσή μας, ε, στην Λιβερία, γύρω 45% της γης ε, έχει δοθεί με συμβόλαια σε ξένους επενδυτές, τα οποία μάλιστα πέρασαν με νόμο το Κοινοβούλιο. Οπότε είναι τα χέρια μας δεμένα. Και όσο σημαντικά και αν είναι τα εθελοντικά πλαίσια και κατευθυντήριες γραμμές, θεωρούμε πως ε, το και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την ε, δύναμη και την ευθύνη να διασφαλίσει ότι θα πρέπει η χρηματοδοτικοί οργανισμοί να τηρούν κάποιου κανόνε. Η Ευρώπη είναι στην πρώτη γραμμή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουν τη μοναδική αυτή ευκαιρία να βοηθήσουν ε, κάποιε από αυτές τις κοινότητε που παλεύουν για να μπορέσουν να αντισταθούν σε αυτές τις δυσκολίες και τους εκτοπισμούς. Σας ευχαριστώ τηρήσατε το χρόνο σας και γιατί είπατε τόσα πολλά σε τόσα λίγα λεπτά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, σημερινούς ομιλητές. Η στιγμή ήταν ε, κέρια, ιδιαίτερα μετά από το ψήφισμα που εγκρίναμε στην Ολομέλεια. Το Κοινοβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα και θέλω να ευχαριστήσω και τους πρέσβεις καθώς και την Εξωτερική Υπηρεσία Δράσης και την Κομισιόν για την ενημέρωση και την πλήρη στήριξη που προσφέρουν καθώς και να ευχαριστήσω τους ε, πολυάριθμους ευρωβουλευτές που ήταν παρόντες σήμερα και ε, μπορείτε πάντοτε να βασίζεστε εδώ σε εμά, σε αυτή την Επιτροπή, αλλά και σε ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ επίσης όλους τους οργανισμούς που εσεί αντιπροσωπεύετε και να σας πω ότι υπάρχει σίγουρη και αποφασιστική δέσμευση και διαμφισβήτητη δέσμευση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευρά μα. Σα ευχαριστώ όλους πολύ. Παρακαλώ να συνεχίσετε τις συζητήσεις εκτός της αίθουσας, γιατί εδώ πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Κυρία Αντιπρόεδρε Λουνατσέκα, μήπως μπορείτε να μετακινηθείτε με το πηγαδάκι σας εκτός, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την ευθύνη των εταιριών και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, πάντοτε δηλαδή στο ίδιο θέμα, εταιρείε και ανθρώπινα δικαιώματα. Για θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεση που ονομάζεται Εταιρική Ευθύνη και Σοβαρές Παραβιάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε Τρίτες Χώρες. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ την υποεπιτροπή μας. Ο εισηγητής είναι ο Ιγνάτσιο Κοράου από το κίνημα Πέντε Αστέρες και την ομάδα EFDD. Και είχε κάνει εξαιρετικά περιστατωμένη δουλειά. Ε, είναι μια προσέγγιση ανοιχτή και το κείμενο δηλαδή καλεί να δράσουμε σε διάφορα επίπεδα για να ρυθμιστούν νομικού τύπου θέματα που προκύπτουν από τον πολυεθνικό χαρακτήρα των εταιριών αυτών. Είναι πραγματική πρόκληση αυτό και στη συνέχεια μιλά για αβεβαιότητες σε σχέση με την ευθύνη ε, για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται ακριβώς άμεσα με τη δραστηριότητα αυτών των εταιριών. Αυτό που μπορώ να προσθέσω είναι ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η Παρασκευή, σε δύο μέρες δηλαδή το μεσημέρι της Παρασκευής και θα συζητήσουμε αυτές τις τροπολογίες στις 30 Μαΐου. Και τώρα φυσικά δίνω μέσα στο λόγο στον Ινάτσιο Κοράο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την εκτιμησή μου και τις ευχαριστίες μου σε όσους συμμετείχαν με την... συμμετείχαν στη διαδικασία και βρίσκονται εδώ σήμερα για να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Μετά από μήνες ακροάσεων, συνεννοήσεων με άλλους ευρωβουλευτές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, Έχω επιτέλους την τιμή να μοιραστώ μαζί σας το πρώτο σχέδιο της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας της εταιρική ευθύνης για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. Πρόκειται για το αποτέλεσμα συνεργασίας και ελπίζω ότι συμπεριέλαβα τις βασικές προτάσεις των διαφόρων συνάδελφων. Θεωρώ πως για να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή έκθεση η συνεργασία όλων των μελών της Προεπιτροπής έχει μεγάλη σημασία. Μάλιστα θεωρώ πως είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα για διάφορα θέματα που αποσχολούν την Επιτροπή μας δικαιώματα εργαζομένων, υποχρέωση των κρατών να προστατεύουν του εργαζόμενου, προστασία του περιβάλλοντος, δικαιώματα αυτοχθόνων πληθυσμών, δικαιώματα των παιδιών κτλ. Είναι γνωστό πόσο ευρύ είναι το φάσμα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ξεκινάει από την απληστία των επιχειρήσεων και η πρόσφατη ιστορία μας δείχνει πόσο συχνά εμπλέκονται οι επιχειρήσεις σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρώτη συνεδρίαση με τους σκιώδεις εισηγητές ε, εστιάστηκε στο να ακούσουμε τις απόψεις και τις ιδέες άλλων ομάδων. Γνωρίζοντας την εξαιρετική σημασία των συνεισφορών των ε, συναδέλφων. Ήταν μεγάλη μου χαρά το ότι διαπίστωσα ότι ε, έχουμε κάποιες κοινέ θέσεις και αρχές. Ε, τη σημασία δηλαδή του θέματος, την ανάγκη άμεσης παρέμβασης, την ε, μεγάλη σημασία του θέματος, ε, το οποίο δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλη μια ωραία αλλά άχρηστη δήλωση, αλλά με τρόπο συγκεκριμένο έχει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό μέσο και βεβαίω τη χρησιμότητα της αυτοδέσμευσης των επιχειρήσεων. Στο ίδιο πνεύμα αποφασίσαμε να αφιερώσουμε τη δεύτερη συνάντησή μας στην ακρόαση των ΜΚΟ της Κοινωνίας των Πολιτών και διεθνών οργανισμών που ειδικεύονται στο θέμα. Στις 13 Ιανουαρίου συναντηθήκαμε ξανά με εκπρόσωπο του υπατορμοστή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα μαζί με αρκετές ε, ΜΚΟ. Μετά στις 28 Ιανουαρίου στο ίδιο πνεύμα συζητήσαμε με ΜΚΟ στο πλαίσιο της συζήτησης ε, ευρωβουλευτών ε, και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση της πολιτικής διαδικασίας για να δώσουμε όθηση στην διαδικασία της δέουσας επιμέλειας. Επίσης, προσπαθήσαμε ακριβώ να λάβουμε υπόψη τι απόψει των ΜΚΟ και να εμπαθύνουμε ορισμένε πτυχέ. Βλέπουμε λοιπόν το αποτέλεσμα όλη αυτή τη διαδικασία σήμερα, η οποία είναι δομημένη στου εξή. Οι επιχειρήσει και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνέ πλαίσιο και εκκλήσει προ τι εταιρείε και η υποχρέωσή του. σέβονται, η υποχρέωση των κρατών μελών ε, να προστατεύουν και βεβαίως οι εκκλήσεις προς την Κομισιόν. Βλέπουμε λοιπόν πως η βασική ιδέα ήταν όχι μόνο να κάνουμε διακηρύξεις παλαιών και νέων δικαιωμάτων, είναι ήδη γνωστά, παρόλα αυτά παραβιάζονται από κάποιες εταιρείες σε τρίτες χώρες. Στόχος μας ήταν να προτείνουμε μέσω της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας πολύ συγκεκριμένα μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση ακολουθώντας μια πάρα πολύ συγκεκριμένη προστασία αυτών των δικαιωμάτων και σε τρίτες χώρες όταν ε, υπάρχουν φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να παρακινήσουμε τις εταιρείε να σέβονται την ομοθεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων εθελοντικά και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ελέγχου Υπό αυτή την έννοια, η παράγραφος 31 ε, που ζητάει την ε, δράση των εταιριών χωρίς ε, παραβιάσεις και οι, οι επόμενες παράγραφοι που ζητούν να υπάρξει δυνατότητα προσφυγής και επανόρθωσης αστικής και ποινική. Κάθε παράγραφος αυτής Τη έκθεση πάει σε αυτή την ε, κατεύθυνση, καθώς λέει πω υπάρχει υποχρέωση των εταιριών να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποχρέωση των κρατών να τα προστατεύουν τουλάχιστον για όσους βρίσκονται εντός της ε, δικαιοδοσίας τους. Γνωρίζω τις απόψεις των πολιτικών ομάδων και καταλαβαίνω πως δεν μπορεί όλοι να δείχνουν όλες τις ε, παραγράφους, αλλά είμαι σίγουρος πως θα καταφέρουμε να ψηφίσουμε την έκθεσή μας τον ε, Ιούνιο με συμφωνία όλων των πολιτικών ομάδων και έτσι η υποεπιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να συνεισφέρει στην ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα τόσο σημαντικό τομέα. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ απεριορίστος κύριε Σιγητά. Ο κύριος Αντρέι Ξύμπ από πλευρά του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, είχαμε κάποιες ε, λεπτομερίες για ένα πολύ δύσκολο ε, θέμα το οποίο αφορά την ευθύνη των εταιριών για ε, σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εδώ λοιπόν θα πρέπει να βρούμε κάποιες ε, συμβιβαστικές να τις ταυτοποιήσουμε και δεν είναι το πρώτο έγγραφο το οποίο αναφέρεται στο συγκεκριμένο ζήτημα, δεν είναι το πρώτο έγγραφο το οποίο συζητούμε εδώ στο Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Όλα τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της θα πρέπει να τηρούν τις ε, δεσμεύσεις τους και τις αξίες τους, όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η οικονομική δραστηριότητα δεν συμβαίνει στο κενό, συμβαίνει στο πλαίσιο συγκεκριμένων συνθήκων και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει πολύ υψηλό παγκόσμιος ανταγωνισμός, ε, υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις ε, και απαιτείται δικαιοσύνη και πρόληψη. Δικαιοσύνη όταν ταυτοποιούμε αυτή την παραβίαση αυτή η γνωμοδότηση για τη δημιουργία νέων συνθήκων και βαρών ε, θα απέναντι σε εταιρείε οι οποίε δεν έχουν κάνει κάποια περιβίωση θα είναι κάτι το άδικο, διότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πηγή υπερνομοθέτησης, ε, ιδιαίτερως όσον αφορά οικονομικές υποθέσεις. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη μία πλευρά και από την άλλη να αποφύγουμε υπερβολικούς κανονισμούς ε, και να δημιουργήσουμε υπερβολικό βάρος. Σε περίπτωση που έχουμε κάτι τέτοιο, τότε υπάρχει η τάση διαρροής οικονομικής δραστηριότητας ε, να πηγαίνουν δηλαδή σε άλλες περιοχές όπου τα στάνταρ είναι χαμηλότερα και αυτό το βλέπουμε για παράδειγμα στον τομέα των κλιματικών αλλαγών και την ομοθεσία που σχετίζεται με αυτό το θέμα. Αυστηροί κανονισμοί ε, όσον αφορά ε, την διανομή αδειών για το διοξίδιο του άνθρακα αυτό οδηγεί σε διαρροές θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει και μια ιδιαίτερη κατηγορία επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις ε, και έχουν διαφορετικές ε, δυνατότητες από τους μεγάλους παίκτες θα πρέπει να τις περιλάβουμε και αυτές λοιπόν και αναφέρθηκε ήδη από σε δύο προηγούμενες γνωμοδοτήσεις του 13 αλλά και μια πρόταση ψηφίσματος που αφορούσε την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την οικονομική δραστηριότητα και την ε, δημιουργία ανάπτυξης ε, και εκεί είχαμε το άρθρο 79 ε, όπου ε, συμφωνήθηκε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια ενιαία προσέγγιση για αυτό διότι υπάρχει μια, αρχική, ε, μια ε, συγκεκριμένη αρχή και ότι, το, ότι ένας κανονισμός μπορεί να ισχύει σε όλα. Θα πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε μια ευελιξία όταν αφαρμόζουμε τις βασικές αρχές και να θυμόμαστε ε, τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα κράτη-μέλη και να λαμβάνουμε υπόψη μας επίσης τις δυνατότητες ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, και στην δεύτερη πρόταση σχετικά με την, με εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη λογοδοσία αλλά και την ε, διαφάνεια των επιχειρήσεων στο άρθρο 39 εκεί πέρα αναφέρεται μια επενθύμηση για το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο σε συγκεκριμένους τομείς και όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ε, το ψήφισμά μας υπενθυμίζει ότι όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχει μια γενικότερη αρχή που λέει ότι αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούν με βάση την αρχή σκέψου ε, περιορισμένα στην αρχή ε, και έχουμε αυτή την προσέγγιση απέναντι στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, διότι οι επιχειρήσεις αυτές πολλές φορές λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο. Ξέρω ότι πρέπει να είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε. Κλείνοντας λοιπόν, είναι σημαντικό να αναπτύξουμε, να δημιουργήσουμε ε, κανονισμούς λαμβάνοντας υπόψη μας όμως το επιχειρησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις και θα πρέπει να το κάνουμε αυτό και σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω του ΟΑΣΑ, ε, του ΟΗΕ ε, μια πρωτοβουλία λοιπόν η οποία θα αυξήσει την διαφάνεια είναι κάτι το οποίο εμείς ε, χαιρετίζουμε, θα πρέπει να την, να την υποστηρίξουμε και θα πρέπει να υπάρχουν και επιστοποιήσεις. Έχουμε για παράδειγμα το ISO αλλά και άλλα πρότυμα. Το άρθρο 26, εδώ έχω κάποια ανησυχία, ε, το οποίο μιλά για την διεύρυνση της δικαιοδοσίας με βάση τον κανονισμό Βρυξέλλες 1 θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τη συνεργασία με την Επιτροπή ε, Τζούρι ε, και αυτό δεν περιλαμβάνεται εδώ. Η ε, γνωμοδότηση από την πλευρά της Τζούρι θα είναι αναγκαία διότι έχουμε να κάνουμε για ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον κανονισμό Βρυξέλλες 1 και το εμπορικό δίκαιο ενώ για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλούμε για ποινικό δίκαιο και θα πρέπει να υπάρχει κάποια αντίδραση ε, που να σχετίζεται με το ποινικό ε, δίκαιο. Ε, εάν θα πρέπει λοιπόν να διευρύνουμε τη δικαιοδοσία, αν αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να επιβάλλουμε τις νομικές μας λύσεις σε άλλες δικαιοδοσίες και σε τρίτες χώρες. Και αν θέλουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί πάνω σε αυτό το ζήτημα και να βασιζόμαστε σε μια καλή συνεργασία μεταξύ των χωρών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φρανσίσκο Ασίσκη, των Σοσιαλιστών. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ξεκινήσω χαιρετίζοντα ε, και πενώντας τον κύριο Γνώσια Κοράου για την ποιότητα της, ε, του σχεδίου έκθεσης που μας ε, υπέβαλε και την μεθοδολογία που χρησιμοποίησε για να κάνει την έκθεση. Πρόκειται για ένα θέμα πολύ περίπλοκο και ευαίσθητο για πολλούς και διάφορους λόγους. Ε, μία από τις πιο γνωστές είναι ακριβώς η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή η δυνατότητα των εταιριών να κινητοποιούνται, να κινούνται ε, αναζητώντας ε, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Δεν είναι νέο το φαινόμενο, όμως αυτό το φαινόμενο έχει πλέον πάρει διαστάσεις τεράστιες, ε, άνευ προηγουμένου. Γι' αυτό και Πρέπει με μεγαλύτερη υπευθυνότητα να το αντιμετωπίσουμε. Στην περίπτωση των ευρωπαϊκών εταιριών αυτή η αύξηση ευθύνη ε, ε, έχει να κάνει ε, με τις αξίες τι οποίες εμεί υποστηρίζουμε. Οι συνέπειε των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στις διάφορε χώρε. πολλές φορέ επηρεάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και μπορεί να είναι καταστροφικέ σε σχέση με τι μειονότητε. Ε, παιδιά και άλλες ευάλωτες ε, μερίδες του πληθυσμού. Πολλές ε, τέτοιες επιχειρήσεις έχουν θηγατρικές ή ευρωπαϊκές ή είναι ευρωπαϊκές. Και γι' αυτό το έγγραφο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ επικοδομητικό. Αναγνωρίζει κάποιε πρόοδου που έχουν σημειωθεί και διάφορα μέτρα έχει υποβάλει, έχει θυσπίσει μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω ο μηχανισμό GSP-SYN. Αλλά όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ε, θα πρέπει να έχουν ε, ελεγκτικούς μηχανισμούς για να ελέγχουν τη δράση των επιχειρήσεών τους σε ξένες χώρες ε, και κατά πόσο οι εταιρείε τους στηρίζουν τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει και δεσμευτική συνθήκη που διαπραγματευόμαστε σε επίπεδο του ΙΕ ώστε να υπάρχει ευθύνη ακόμα και ποινική των εταιριών όταν αυτές προβαίνουν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια από τις πιο ζωντανές συζητήσεις σε αυτό το τομέα και τις πιο δύσκολες συζητήσεις είναι να γνωρίζουμε πώς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δουν αν και να δουν και να ελέγξουν πώς και αν οι εταιρείε τους ε, διαπράττουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν αυτές εγκαθίστανται σε τρίτες χώρες όπου δηλαδή εμείς δεν έχουμε δικαιοδοσία. Ε, Φόρανε σε ε, Πρέπει να μπορούμε να εντοπίσουμε και σε ομάδες τρίτων χωρών και να μπορούν οι χώρε, ή μάλλον οι αδικημένοι να καταφύγουν και στη δικαιοσύνη των κρατών μελών. Αυτή είναι μια λύση που προτείνει αυτή η έκθεση. Γι' αυτό και εν γέννη είμαστε σύμφωνοι με αυτή την έκθεση. Θα υποβάλουμε κάποιες μικρές τροπολογίες που θέλουν να αποσαφηνίσουν περισσότερο κάποιες διατυπώσεις και θα συγκεκριμενοποιήσουν κάποιες ιδέες από αυτές που υπάρχουν εδώ σε αυτή την έκθεση, όπως τη δυνατότητα να, μελετηθεί το ενδεχόμενο να ε, μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε μια ευρεία εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού, ώστε να προτιμά προϊόντα από εταιρείε που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στι τρίτε χώρε. Πάντω, για να κλείσω, θέλω να πω κατ' ουσίαν ότι πρόκειται για μια έκθεση όπου ε, συμφωνούμε γιατί τοποθετεί τα θέματα πολύ καλά, με ισορροπία, αλλά και ταυτόχρονα με τη φιλοδοξία να αλλάξουν κάποια πράγματα για να λυθούν αυτού του τύπου τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από την ομάδα των συντηρητικών, ο κ. Άρνε Κέρικε. Ευχαριστώ πολύ για τη συγκεκριμένη έκθεση. Όσον, αφορού, όταν αφορά την Ευρώπη, θα πρέπει να εξετάσουμε τις δικές μας αξίες, ε, οι οποίες θα πρέπει να είναι το σημαντικότερο εξαγωγικό προϊόν μας. Μιλάμε για τα ευρωπαϊκά ε, ιδεώδη του ε, τίμιου εμπόρου όταν ε, το θέμα αφορά ευαίσθητα ζητήματα όπως αυτό στην έκθεση όσον αφορά την ευθύνη των επιχειρήσεων για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. Κατά την εφαρμογή αυτού δεν μπορούμε να μιλάμε για επιχειρήσεις και για ανθρώπους πρώτης ή δεύτερης ε, τάξης. Χαιρετίζω την έκθεση και συγκεκριμένα κάποια σημεία. Για παράδειγμα, αναφέρει στη βασική αρχή των Ηνωμένων Εθνών ε, για την οικονομία και τα ανθρωπίνα δικαιώματα η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες που διαπράττονται ε, από επιχειρήσεις είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα ε, και αυτό φαίνεται και στις αναφορές ε, της εταιρικής κοινωνικής ε, ευθύνης. Χαιρετίζω θα ήθελα να αναφερθώ στην αναφορά του ΟΗΕ για τον ρόλο των επιχειρήσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους αυτό στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βέμπα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τα όσα είπε. Μόλις είχαμε μια ακρόαση που συσχετιζόταν με το θέμα, οπότε σίγουρα είχαμε την ευκαιρία να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα την διάσταση των, παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει ε, να ε, απευθυνθούμε με το σωστό τρόπο σε αυτό το φαινόμενο. Έχω οριζε, ορισμένα ερωτήματα όμως προς τον εισηγητή για να καταλάβω καλύτερα τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε και, ποια, και τι είδους εργαλεία θέλετε να έχουμε. Αρχικά, αν μου επιτρέπετε, παρατήρησα μία ε, αντιπαράθεση στην παράγραφο 6 όπου λέτε ότι πρέπει να υπάρχει νομική υποχρέωση για την αποφυγή ε, παραβίωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, ε, σε κάποιο άλλο σημείο όμως λέτε ότι θα πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικά μέτρα και το βασικό μου ερώτημα λοιπόν σχετικά με τις προτάσεις που κάνατε στην παράγραφο 10 για παράδειγμα, 12, 18 σχετίζονται με το ζήτημα της δικαιοδοσίας. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζουμε το συγκεκριμένο θέμα, διότι μου φαίνεται ότι είναι δύσκολο ε, κάνουμε πιο δύσκολο τον νομικό τρόπο σκέψης προσωπικά δεν καταλαβαίνω το πώς ο κανονισμός Βρυξέλλες 1 μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτά τα οποία προτείνεται. Θα έπρεπε λοιπόν να, θε, να θέσουμε ένα ερώτημα στην νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, διότι πρέπει να έχουμε κάτι το οποίο είναι ακριβές και μπορεί να εφαρμοστεί. Έχω μία ερώτηση σχετικά με το άρθρο 19 όπου αναφέρατε μηχανισμούς ε, ε, συλλογικής ε, προσφυγής και στη συνέχεια στο 22 ζητάτε δεσμευτικούς κανονισμούς και μηχανισμούς ανεξάρτητης παρατήρησης και πάλι θέλω να το εξηγήσετε καλύτερα στην ε, έκθεσή σας έχετε περιορισμένη έκταση των όσων μπορείτε να πείτε, όμως θα ήθελα να γίνετε ε, πιο συγκεκριμένους σε αυτά που αναφέρεστε. Και τέλος, θέλω να καταλάβω καλύτερα το φόρουμ να της, διότι ε, λέτε ότι αυτό το φόρουμ θα πρέπει να παίζει ένα ρόλο στους τομείς που επηρεάζονται δεν αναφέρεστε σε μια ε, νομική ε, δράση, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω τι ρόλο θα παίξει. και θα ήθελα να σημειώσω μία ε, αντίφαση στην παράγραφο 1 μιλάτε για τέτοια προϊόντα και ότι θα πρέπει να είναι σε θελοντική βάση και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ θα υποστήριζα. Στο τέλος όμως αναφέρεται ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σώμα το οποίο θα επικυρώνει ε, και θα πιστοποιεί κάτι τέτοιο. Αυτό εμένα μπερδεύει διότι άμα είναι σε εθελοντική βάση τότε δεν έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε την ανάγκη ενός τέτοιου ε, σώματος. Θα ακούσω τις απαντήσεις σας και μετά θα ξέρω πώς να συνεχίσω με τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ εξ ονόματος των Πρασίνων, η κυρία Νόχμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο δικός μας ως κοιόδης ηγητής, ο κύριος Κλάους Μπουκνερ, δυστυχώς απουσιάζει, οπότε θα σας ε, πω σύντομα το μήνυμά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γνάσιο Κορέο για το πολύ καλό σχέδιο έκθεσης και για την ακρόαση που οργανώσατε με τις ειδικέ ΜΚΟ και λάβαμε έτσι αρκετές καλές ιδέες. Θεωρούμε πως οι προηγούμενες εκθέσεις που ασχολήθηκαν με την εταιρική κοινωνική ευθύνη συμπληρώνονται πάρα πολύ καλά με την δική σας έκθεση και αναφέρομαι στην ακρόαση που είχαμε μόλις και για τα δικαιώματα της γης ότι δεν μπορεί να μιλάμε μόνο όταν μιλάμε για προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων για εταιρική κοινωνική ευθύνη. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο το οποίο θα δεσμεύει νομικά τις ε, εταιρείες. Και έτσι οι δικές μας οι τροπολογίες που θα τις ε, στείλουμε αύριο θα πηγαίνουν προς αυτή την ε, κατεύθυνση που πάει και η έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Για την άκρα αριστερά, ο Μιγγέλ Ούρμπαν Κρέσπο. Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να καταρχάς να σχολιάσω και να χαιρετήσω την πρωτοβουλία του συναδέλφου Κοράου. Ε, τη θεωρούμε πολύ απαραίτητη και, απαραίτητη και επίγουσα πριν να, να καταρχάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις κακές πρακτικές από πλευράς ευρωπαϊκών εταιριών στις τρίτες χώρες. Ευχαριστώ για τη δουλειά σας και για την πρωτοβουλία. Η πολίτικα διαπραγματεύσεων για εμπορικές συμφωνίες που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες οι επιχειρήσεις λειτουργώντας σε τρίτες χώρες όπου δεν υπάρχουν επαρκείς εγγύησεις ώστε να ε, ενημερώνεται και να εμποδίζει η Κομισιόν ε, την διάπραξη παρανόμων ε, δράσεων είναι προφανέ. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν μηχανισμοί ώστε να εξασφαλιστεί η αστική και η ποινική ευθύνη ενώπιον των δικαστηρίων του κράτου προέλευση τη κύρια εταιρεία, τη μητρική εταιρεία, όταν διαπιστώνονται παραβιάζει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γι' αυτό θα καταθέσουμε μια σειρά τροπολογίε που συμφωνούν με την αρχική πρόταση και λίγο πιο πέρα. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να, ε, να ζητήσουμε τη δημιουργία δεσμευτικών μηχανισμών. Αυτό είναι θεμελιώδη σημασία γιατί είναι απαραίτητο οι επιχειρήσει να λογοδοτούν αστικά και ποινικά ενώπιον του κράτου προέλευση τη επιχείρηση, σε αυτή την περίπτωση την Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκά κράτη, όσον αφορά τι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. τη ρήτρε προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολύ συχνά αναφερόμαστε σε αυτέ και μιλάμε για αυτέ, αλλά νομίζουμε ότι θα είναι αποτελεσματικέ μόνο αν συνδεθούν με δεσμευτικού μηχανισμού που θα προβλέπουν και οι και αποζημιώσει. Διότι διαφορετικά θα συμβαίνει ότι, ότι συνέβαινε ανέκαθεν, δηλαδή ψηλά γράμματα. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργηθεί ένας δημόσιος οργανισμός για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών εταιριών στα τρίτε χώρες και μάλιστα να μπορούν να ακυρωθούν αυτές οι πρακτικές και να λογοδοτούν ανάμεσα σε άλλα θεσμού και σε αυτό το κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να παρακολουθούμε την ε, υλοποίηση αυτής της ρήτρα και την τήρηση της. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω πως με τόσες δεσμεύσεις δεν θα πνίξουμε την οικονομία. Γιατί αν φανταζόμαστε η οικονομία είναι μόνο κάτι το οποίο πρέπει να ελέγχεται, ε, θα, απο, θα αποθάνει. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Όχι, δεν θέλει κανείς να καταστρέψει καμιά οικονομία. Ναι, καμιά φορά χωρίς να το θέλουμε το κάνουμε εάν λάβουμε λάθος αποφάσεις. Ναι, μα... Ναι, Όταν εσείς ο ίδιος μιλάτε για ακροαριστερά, ε, ενώ να λέτε νοτική αριστερά, ήδη ε, θέλετε να προκαθορίσετε αυτά που λέω. Όχι, εντάξει, ήταν μια σύντομη παρατήρηση. Σας ευχαριστώ για την ε, προσοχή σας. Ο κύριος Χρήστο τώρα από πλευρά των σοσιαλιστών. <coughs> Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο μίλησε για την, την έκθεση. Εγώ θέλω να μιλήσω για την επόμενη. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Θα ακούσουμε τώρα τον αρμόδιο από την ε, Κομισιόν, τον κύριο Ρικάρντο Σέρι. Έχει το λόγο παραπαλώ όμως σύντομα. Ναι, θα είμαι πολύ σύντομος. θα ήθελα εξ ονόματος υπηρεσίας εξωτερικής δράσης να επενέσω αυτή την έκθεση όπως είπε ο κύριος Κοράο ε, έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά και διαβουλεύσεις γιατί βεβαίως είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση, εστιάζει στα κυριότερα ζητήματα και στηρίζει βεβαίως τα όσα υπόθηκαν και από άλλους βουλευτές, γιατί αυτό το οποίο προκύπτει είναι πως ε, είναι, θα έλεγα, πολύ σωστά δομημένη και ισορροπημένη η έκθεση. Είναι ένα θέμα αρκετά επίμαχο. Νομίζω όμως πως υπάρχουν αρκετές προτάσεις οι οποίες ε, έχουν ε, βεβαίως μεγάλη σημασία και είναι ενδιαφέρουσες. Ε, η υπηρεσία μας βεβαίως δεν είναι ακριβώς αρμόδια. Όπως λέει και η έκθεση πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει διάφορες νομικές και πολιτικές πτυχές και οπωσδήποτε αφορά και εμάς αλλά και άλλους συναδέλφους και διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε δεν θα απαντήσω εγώ σε όλες τις προτάσεις σας. Θα πω όμως πως σε γενικές γραμμές είναι κάτι το χρήσιμο, το επίκαιρο. Νομίζω πως ε, είναι σημαντικό να ξαναδούμε τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα, όπως είπε η κυρία Λοχπίλερ, και το θέμα της αρπαγής γης σχετίζεται με αυτή την έκθεση και είχα την ευκαιρία να πω το τι κάνουμε σε αυτόν τον τομέα, να υπενθυμίσω τώρα το χρονοδιάγραμμα. Έρχεται την κατάλληλη στιγμή γιατί θα θυμάστε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται ένα νέο έγγραφο πολιτικής ε, θα λέγαμε για την ε, εταιρική κοινωνική ευθύνη που ελπίζουμε να είναι έτοιμο μετά το καλοκαίρι αλλά υπάρχουν δύο παράλληλα σχέδια συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Το ένα αφορά υπεύθυνη παγκόσμια αλυσίδα προσθέμενης αξίας και το άλλο φορά ακριβώς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε δεν έχουμε όλα αυτά τα θέματα της δεσμεύσης αλλά και την ε, εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω πως και η έκθεσή σας εδώ πέρα θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ακριβώς ε, για να κάνει προτάσεις. Τέλος, μου επιτρέπετε για τον δεσμευτικό ή μη χαρακτήρα, να επαναλάβω την θέση μας. Οι συνάδελφοι ίσως από την Κομισιόν είναι σε καλύτερη θέση να περιγράψουν την θέση τους, αλλά σε γενικές γραμμές από το 2011 το σκεπτικό μας είναι πως το θέμα αυτό πρέπει να το δούμε με ένα μείγμα δεσμευτικών και μη δεσμευτικών μέσων. Αναφέρατε, παραδείγματο χάρη, την οδηγία για την μη αποκάλυψη οικονομικών στοιχείων είναι δεσμευτική και ανταποκρίνεται σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται κάποια δεσμευτική προσέγγιση. Για την συνθήκη τώρα, ε, κάτι το οποίο μας αφορά περισσότερο, για ένα νομικά δεσμευτικό μέσο το οποίο συζητιέται στην Γενέβη, αυτό βέβαια θα απαιτήσει αρκετές συζητήσεις, αλλά σε γενικές γραμμές για να συνοψίσω η θέση της Ένωσης είναι ότι δεν έχουμε ενεργό εμπλοκή στην ομάδα αυτή με βάση δύο κύριος αιτήματα που έγιναν. Πρώτον, ότι δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε τις κατευθυντήριες αρχές που υπάρχουν και το σημαντικότερο το γεγονός πως το πεδίο εφαρμογής ε, του νομικά δεσμευτικού μέτρου θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τις πολυεθνικές αλλά και τις τοπικές εταιρείες που συχνά είναι υπεύθυνε για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν ε, έχει γίνει ακόμα δεκτή στην Γενέβη αυτή η πρόταση, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να επιμείνουμε, όπως και πολλές ΜΚΟ. Ελπίζουμε λοιπόν, αν πάμε σε μια πιο ενεργό εμπλοκή να γίνουν αυτά δεκτά. Σας ευχαριστώ. Σύντομες απαντήσεις από τον εισηγητή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ε, από την εξή ε, προϋπόθεση. Γνωρίζουμε ότι το θέμα είναι περίπλοκο και δύσκολο. Πρέπει να κατανοήσουμε τι στόχο έχουμε ως Επιτροπή, Υποεπιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ως Ευρωκοινοβούλιο. Ε, ως Υποεπιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, θέλουμε να καταλήξουμε σε μια ισχυρή θέση κατά τη γνώμη μου, ενισχυτική ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα για τον έλεγχο και για τις κυρώσεις και ε, τις καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευρά των πολυεθνικών. Τώρα από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει να κάνει με την ΑΦΕΤ και με την Ολομέλεια, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ορίσουμε έναν βελτιωτικό τρόπο όσον αφορά την, το διεθνή ανταγωνισμό. Δηλαδή, ο διεθνή ανταγωνισμό μπορεί να οδηγεί στο ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα είναι χαμηλότερος, χαμηλότερη. Εμεί πρέπει να δημιουργήσουμε το κίνητρο και για του άλλου ώστε να βελτιωθούν. Έπειτα, η το βασικό όμω σχέδιο έκθεση που έγινε σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον κανονισμό δεν μπορούσε να τα περιλαμβάνει όλα και γι' αυτό και πολλέ από τι παρατηρήσει που θα προέλθουν από τι ομάδε θα αποτελέσουν τμήμα τη τελική έκθεση γιατί ε, θα ψηφιστούν στο τέλο. Και αυτό για να πω ότι συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπατε, πολλέ από τι παρατηρήσει ε, των συναδέλφων όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την πρόληψη και κυρίως για να μην δημιουργηθούν ε, επιβαρύνσεις ε, ε, μεγάλες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε κανένας να καταστρέψει την οικονομία όπως είπε ο κύριος Πρέντα. μετά από την παρέμβαση του Ρουμπάνου. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας, όχι. Θέλουμε να αυξήσουμε το επίπεδο προστασίας, να μην συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Γνωρίζουμε ο ότι η Προεδρία η Ολλανδική είναι πέρα αυτή τη προσέγγιση, αλλά θέλουμε βεβαίω να μπορούν να δουλέψουν οι επιχειρήσει μα Να απαντήσω σε κάποιε ερωτήσει. Η άποψη τη δικαιοδοσία βέβαια είναι ε, δύσκολη. Είναι δύσκολο να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα δικαιοδοσία εν γέννη μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και σαφώ είναι ακόμη πιο περίπλοκο όταν μιλάμε με χώρε εκτό. Όμω η ευθύνη που μπορεί αυτή τη στιγμή να μας βαραίνει λόγω της λειτουργίας της ε, δικαιοδοτικής και αν σύνδεται μόνο με το, η χώρα προέλευση τη εταιρεία είναι κάτι το οποίο εμεί μπορούμε να ζητήσουμε. Δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί δεν έχουμε τέτοιου είδου αρμοδιότητα. Δεν έχουμε τέτοιο σύστημα δικαιοδοσία για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω μια πρόταση μπορούμε να την κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά για το φόρουμ νεσισιτάτης, που είναι ένας όρος που μάθαμε από το Πανεπιστήμιο, αναφερόμαστε στη δυνατότητα να ζητήσουμε τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη στο δικαιοδοτικό σύστημα ενός κράτους τη δυνατότητα ένα άλλο να μπορέσει να, ε, να καταφύγει στο σύστημα που το, το καλύπτει. Αν ας πούμε το γαλλικό σύστημα ε, αντί το λετωνικό προβλέπει περισσότερη προστασία ή περισσότερη πρόσβαση στα μέσα της δικαιοσύνης, τότε θα πρέπει να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στο γαλλικό σύστημα δικαιοσύνης. Έπειτα μιλάμε για cross-section και συλλογική προσφυγή για περίπτωση δηλαδή ε, παραβιάσεων που αφορούν πολύ κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Για τι πράγμα, για εκμετάλλευση δαφών, γεών, υπόρων. Όταν μιλάμε για το σήμα abuse free με όλες τις δυσκολίες όσον αφορά ε, τη δυνατότητα εφαρμογής και ελέγχου δεν είναι αντίφαση. Σαφώς υπάρχει εθελοντική βάση. Υπάρχει εθελοντική βάση να θέλει κανείς δηλαδή να τοποθετήσει αυτό το σήμα. Δεν το βάζουν ωστόσο όλοι και κανένας δεν ελέγχει. Δηλαδή θα πρέπει να προβλεφθεί ένας μηχανισμός ελέγχου στο εσωτερικό της Κομισιόν ή μέσω κάποιου οργανισμού της Επιτροπής, αυτό θα χρησιμεύεται στο να καταστεί αποτελεσματική η χρήση ενός τέτοιου σήματος. διαφορετικά θα πάνε να βάλουν όλοι αυτό το σήμα, abuse αλλά κανένας δεν θα ελέγχει. Αν κάνω σε θελαντικά από μόνο του, του κατέβει και λέει ότι εγώ είμαι μια πολυεθνική που εργάζομαι σε αυτέ τι περιοχέ και σέβομαι ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να κάποιο να το ελέγχει αν όντω ισχύει. Επίση, συμφωνώ με τη λογική για τι ευθύνε και για τη συμφωνία που έχει γίνει και εν γέννη θα πρέπει να αναζητήσουμε, γιατί δεν θα είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν ένα σωρό επιχειρήματα που έχουν αναφερθεί και πολλά πράγματα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις τροπολογίες, στις συμβιβασμούς, στις συμβιβαστικές τροπολογίες, δηλαδή στις επόμενες μας συναντήσεις θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο ώστε να καταλήξουμε σε ένα ε, δυνατό κείμενο. Δεν θα αλλάξουμε βέβαια τον κόσμο σε μια μέρα, όπως και η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να κάνουμε ένα βηματάκι, να δείξουμε ότι έχουμε ένα σαφή μακροπρόθεσμο στόχο. Αυτό ελπίζω πως θα είναι αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης από την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Όπως έλεγα, 22 Απριλίου την Παρασκευή είναι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών και θα τη συζητήσουμε στις 30 Μαΐου. Και τώρα, καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων εκτός της Ένωσης ε, είναι εξέταση των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί για αυτή την έκθεση. Έχουμε λάβει 215 τροπολογίες, εκ των οποίων ορισμένε ε, εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων επιτροπών της Επιτροπής Γυναικών και της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό το γεγονός. Υπήρχε συζήτηση ανάμεσα στην Επιτροπή Δικαιωμάτων και Γυναικών και ΛΥΜΠΕ και στη συνέχεια μετά από πολλούς μήνες και μάλιστα διαπραγματεύσεων και σε συνεννόηση με τους εισηγητές αυτών των επιτροπών Αυτές οι τροπολογίες ε, θεωρήθηκαν αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Γυναικών και της Επιτροπής ε, ε, ΛΥΜΠΕ. Για αυτές λοιπόν τις τροπολογίες πρόκειται για τις 5, 14, 28, 32, 45, 48, 55, 58, 106, 108, 122, 124, 128, 135, 136, 137 και 183. Και να είμαι σίγουρος ότι δεν προλάβατε καν να το σημειώσετε, αλλά θα σας το στείλουμε και γραπτός. Και Έπρεπε να σας τις αναφέρω τώρα. Οι άλλες που είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΛΥΜΠΕΙ έχουμε τις τροπολογίες 114, 123, 157, 163, 172, 210 και 215. Αυτές οι τροπολογίες δεν είναι παραδεκτές στην έκθεση της δικής μας Επιτροπής και τώρα δίχως περαιτέρω καθυστέρηση δίνω το λόγο στην κυρία Μπάρμπαρα Μπίλερ Κυρία Ισηγήτρια, έχετε 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ε, και τα εισαγωγικά στο σχόλια ήταν άριστα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδες για την καλή συνεργασία όσον αφορά τις ε, τρομολογίες και είχαμε και μια πολύ επικοδομητική συνεργασία για την εξέβρεση συμβιβαστικών. Χαίρομαι επίσης ε, για το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Ντρουά ε, συζητά το θέμα της εμπορίας ανθρώπων με αποτέλεσμα να ρίχνει φως σε ε, μία από τις ε, πιο ε, κερδοφόρες εγκληματικές δραστηριότητες στον πλανήτη. Όπως ξέρετε η εμπορία ανθρώπων αποτελεί κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραβιάζοντας την αξιοπρέπεια και την φυσική και ηθική ανεξαρτησία των ανθρώπων μετατρέποντάς τους σε ένα προϊόν. Η συγκεκριμένη έκθεση τονίζει την ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να εντατικοποιήσει ε, και να κάνει προτεραιότητα τη μάχη ε, κατά της εμπορίας των ανθρώπων χρησιμοποιώντας κάθε μέσο στη διάθεσή της για να θέσει ένα τέλος σε αυτή τη δραστηριότητα. Όπως είπατε πρόεδρε, έχουμε λάβει 215 τροπολογίες από τις οποίες κατορθώσαμε να έχουμε 28 συμβιβαστικέ και ενσωματώσαμε λοιπόν πάνω από το 1 τρίτο των τροπολογιών. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε ε, πραγματική συζήτηση σχετικά με την πολιτική κατεύθυνση ε, της έκθεσης ε, ούτε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των σκιωδών ούτε και στη συζήτηση για τις τροπολογίες. Αυτό λοιπόν δείχνει τη μεγάλη, τη μεγάλη συμφωνία που έχουμε πάνω στο θέμα ούτω ώστε η εμπορία ανθρώπων να γίνει ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν δύο ε, σχετικές επιτροπές, η ΦΕΜ και η ΛΥΜΠΕ. Ε, η ΦΕΜ ψήφισε στην αρχή της εβδομάδας ε, και η ΛΥΜΠΕ θα ψηφίσει την επερχόμενη εβδομάδα. Τα σημεία του κειμένου τα οποία συντάχθηκαν με αποκλειστική ευθύνη ε, θα συζητηθούν στην Τρουά πριν από την ε, συζήτηση της ΑΒΕΤ στις 23 του μηνός. Αυτά τα οποία έχουν ε, κοινή ευθύνη όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων θα ψηφιστούν την ίδια μέρα. Υπάρχει επίσης μια γνωμοδότηση από την πλευρά της ΕΝΒΗ η οποία υιοθετήθηκε ήδη τον Μάρτιο και η συγκεκριμένη αφορά κυρίως το εμπόριο οργάνων. Για άλλη μια φορά λοιπόν θα ήθελα να, ευχαριστήσω όλους τους ε, σκιώδεις ε, και όλους συμμετείχαν στη διαδικασία για να έχουμε αυτή την έκθεση και ε, χαίρομαι ε, για την ψηφοφορία που θα ακολουθήσει και θα έχουμε την τελική ευελπιστό ψηφοφορία πριν από την διακοπή για το καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ. Η Σκιώδης ε, Κομοντίνη ψηφίζει σε μια άλλη επιτροπή. Μου ζήτησε λοιπόν να σας ευχαριστώ, ευχαριστήσω μόλις, μόλις μπήκε. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Κομοντίνη Κάτσια για δύο-τρία λεπτά. Διότι έχουμε καθυστερήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και... Ταυτόχρονα υπήρχε ε, μία ε, ψηφοφορία στη Γιούρη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις συμβιβαστικές. Νομίζω ότι κάναμε μεγάλη πρόοδο ε, πάνω σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τους Κιώδης ε, και την εισηγήτρια που κατανόησαν τη θέση μας πάνω στις συμβιβαστικές. Ήταν ένα σημαντικό θέμα για εμάς ε, να έχουμε όσο το, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμφωνία πάνω σε αυτό το θέμα και είμαι βέβαιη ότι οι σκιώδεις καταλαβαίνουν ότι η θέση του EPP ε, πάνω στο δεύτερο κομμάτι της συμβιβαστικής. Ε, επίσης υπάρχουν και άλλες τροπολογίες πάνω στις οποίες θα ψηφίσουμε και θα έλεγα ότι υπάρχουν αρκετές τροπολογίες αναφερόμενοι τώρα σε μερικές εξ αυτών από την πλευρά μας είναι σημαντικό οι τροπολογίες που επικεντρώνονται κυρίως σε ευάλωτους ανθρώπους ε, που μπλέκονται στην εμπορία ανθρώπων Καταλαβαίνω προσωπικά ότι όλα τα θύματα εμπορίας είναι ευάλωτα αυτοί άνθρωποι, όμως υπάρχουν ε, συγκεκριμένες κατηγορίες όπως είναι παιδιά καθώς και άνθρωποι με αναπηρίες. Ε, ευελπιστώ να υπάρξει υποστήριξη σε αυτές τις τροπολογίες. Πέραν τούτου πιστεύω ότι η συγκεκριμένη έκθεση ιδιαίτερω με τις ε, συμβιβαστικές που έχουμε επιτύχει θα, θα δεχτεί ε, υποστήριξης και θα ήθελα πάλι να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος ε, Τσέλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα αρχικά να συγχαρώ την εισηγήτρια για το πολύ καλό κείμενο εγώ μαζί με τους συναδέλφους μου ε, προτείναμε κάποιες ε, τροπολογίες για να διευρύνουμε το πλαίσιο ε, της έκθεσης. Επικεντρωνόμαστε σε θέματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως, όπως είναι ο ρόλος των κυβερνήσεων, ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα τα οποία επιτρέπουν την άνθηση της εμπορίας ανθρώπων. Ε, θέλουμε ε, η, οικονομία να, ε, προ, να αναγκάσει τις κυβερνήσεις να θέσουν ξεκάθαρους στόχους όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υιοθέτηση πολιτικών που προωθούν μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη αναφορά σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Όσον αφορά την συνεργασία σε ε, διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, ε, και τέλος η επανενσωμάτωση των θυμάτων στην κοινωνία και το δικαίωμα ε, να υποφελουθούν προστασίας. Θέλουμε να έχουμε μια επικοδομητική, είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο και χαίρομαι για το πνεύμα και το περιεχόμενο των ε, τροπολογιών που συμπεριλαμβάνονται στις συμβιβαστικές θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λόχμπίλα καθώς επίσης και, του και τους συναδέλφους μου σκιώδης ε, για τις ε, συζητήσεις που είχαμε και είμαι πεπισμένος ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό τελικό κείμενο. Η ε, κυρία Λόκμπιλερ συνεισέφερε τα μάλλα στο στο εμπόριο ανθρώπων στην καταπολέμηση ε, της εμπορίας ανθρώπων. Και πιστεύουμε ότι θα παίξουμε σημαντικό ρόλο πάνω σε αυτό. Στην στρατηγική ε, του 2016 ε, για το αντιτράφικινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Σας ευχαριστώ κύριο Μπασίρ για τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς. Κύριε Πρόεδρε, έχετε κάποιον άλλον αδερφό στην Επιτροπή Ανάπτυξης γιατί είδα κάποιον που σας μοιάζει πολύ. Ωραία, λοιπόν. Συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, την εισηγήτρια και τους και οδησηγητές για την προσέγγιση τους στις διαπραγματεύσεις μέχρι στιγμής. Όπως ξέρετε, το ECR πάντα στηρίζει τον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων και οι βουλευτές μας είχαν εμπλακεί στην σύνταξη της ε, σχετικής οδηγίας. Μάλιστα η κυβέρνησή μας στο Ηνωμένο Βασίλειο επέλεξε να εφαρμόσει αυτή την οδηγία. Υπάρχουν όμως κάποιοι τομείς οι οποίοι είναι προβληματικοί και ανησυχώ ιδιαίτερα για την πίεση που ασκείται στις ευρωπαϊκές εταιρείε που λειτουργούν στο εξωτερικό. Με συγχωρείτε να θυμόμαστε πως σε γενικές γραμμές οι εταιρείε μας προσφέρουν καλύτερες ε, συνθήκες εργασίας από τους εργοδότες της χώρας του τρίτου κόσμου και είναι πιο προσεκτικές όταν μιλάμε για υπεργολαδίες και αγορές πρώτων υλών και προμηθειών. Θεωρώ πως ε, τον αναγκάσουμε τις εταιρείε μας να λογοδοτούν για την ε, εμπορία ανθρώπων οπουδήποτε στην ε, αλυσίδα εφοδιασμού είναι πάρα πολύ αυστηρό. Γι' αυτό ελπίζω η συμβαστική τροπολογία 17 να ψηφιστεί σε μέρη όπως ζήτησαν και άλλες ομάδες. Πέρα από αυτό είμαι ικανοποιημένος με τις υπόλοιπε συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Μία από τις δικές μου τροπολογίες και τρεις ε, του συναδέλφου του κυρίου Τόμα Σέκα από το ECR έχουν συμπεριληφθεί και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους συναδέλφους ε, που βοήθησαν γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους φιλελεύθερους κύριε Βέμπερ. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, να συμφωνήσω και εγώ με τους ε, συναδέλφους που συνεχάρισαν την κυρία Λοχπιλήρ για τη δουλειά που έχει κάνει και για το πνεύμα που επέδειξαν όλοι οι σκιώδεις εισηγητές. Νομίζω πως η έκθεση και οι συμβαστικές ε, τροπολογίες αντικατοπτρίζουν κάποια ζητήματα που όλοι τα έχουμε κατά νου κάποια μέσα για να αντιμετωπίσουμε τις βαθιές αιτίες του φρικτού αυτού φαινομένου. Ε, η άμεση ανάγκη για προγράμματα ενημέρωσης για να μπορεί κάποιος να ταυτοποιεί τα θύματα, η ανάγκη να αναπτυχθούν ε, μέτρα προστασίας των ευπαθών ομάδων, ε, ειδικά των γυναικόπαιδων, ε, μέτρα επανένταξης, πρόσβαση στην δικαιοσύνη, μη ποινικοποίηση, όλα αυτά νομίζω είναι ο πυρήνας αυτής της έκθεσης, αλλά είμαι και πολύ ικανοποιημένη, καθώς κάποια από τα ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την άλλη, την πολιτική μου ομάδα, επίσης έγιναν δεκτά στις συμβιβαστικέ τροπολογίες και τις στηρίζουν και άλλες ομάδες, όπως το θέμα των ανήλικων στρατιωτών, την ανάγκη εξασκησής δέουσας μέλης για να αποφευχθεί η διαφθορά, την ανάγκη να έχουμε κάποιες επενδύσεις σε μηχανισμούς ε, ταυτοποίησης ε, των θυμάτων αυτών ε, μέσα στα κύματα μεταναστών ε, και τούντων άσυλο και καθώς μίλησα και στους συναδέλφους στις Επιτροπές ΛΥΜΠΕ και ΦΑΜ δεν έχω καμία αμφιβολία πως τα όσα ψηφίζουν θα συνεισφέρουν σε αυτή την έκθεσή σας. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για αυτή την συνεργασία. Ευχαριστώ Ιγνάσιο Κοράο για το EFTD. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να μην επαναλάβω πράγματα που έχουν ήδη ακουστεί από τους συναδέλφους. Νομίζω πως το θέμα αυτό σχετίζεται με τα όσα είπαμε πριν, γιατί καμιά φορά μιλάμε για ευρωπαϊκές εταιρείε εκτός ε, της ε, Ευρωπαϊκή Ένωσης, οπότε υπάρχει μια σύνδεση. Και είναι σημαντικό. Ε, και ευχαριστώ την κυρία Λοχμπίλερ για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι στιγμής για να βρει κάποιες συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Νομίζω λοιπόν πως είναι σημαντικό να βρεθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος για να υπάρξουν κυρώσεις γιατί τα νούμερα λένε πως το ποσοστό καταδικών είναι πάρα πολύ χαμηλό. Οπότε ελπίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε κάπως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ζητάει κάποιος άλλος τον λόγο. Κυρία Λόχμπιλερ. Δεν έχω τώρα τίποτα να πω. Θα δω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπασίρ, αν είναι δυνατόν να έχουμε μια χωριστή ψηφοφορία. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω τα, τα είχαμε. Σας ευχαριστώ όλους. Και τώρα περνάμε στο σημείο 11 της ημερής διάταξης, τα... την αναφορά για την αντιπροσωπεία ε, ε, τη επιτροπή μα στη Γενέβη και στη Καμπότζη. Η κυρία Βαλενσιάνο ηγήθηκε τις αποστολές Ξύπ και Μανέσκου Έλκας, για από τους ε, σοσιαλιστές, και συντηρητική, η κυρία Μπεατρίς Μπεσέρα της Άλντε και η κυρία Τζούντιθ Αργεντίνη από τους Πρασίνους πήγαν στη Γενέβη. Η επίσκεψη θα, την αναφορά θα μας κάνει η κυρία Σολέα Πόστ, γιατί η κυρία Βαλενσιάνο λείπει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως βλέπω δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Έχω να δώσω το λόγο ε, και στους συνάδελφους και να μιλήσει σχετικά με την Καμπότζη. Όπως ε, αναφέρατε, όλα τα, όλοι οι ευρωβουλευτές που ήταν μαζί μας ε, στην Κενέβη, ε, ε, έχει γίνει παράδοση να συμμετέχουμε στην συνεδρίαση τους. Ήμασταν 7 μέλη στις 14 και 15 Μαρτίου και εκεί συναντηθήκαμε με ε, ορνομοδότες, με εισηγητές, ε, με τον πρόεδρο, ε, με αξιωματούχους της υπηρεσίας του ΟΗΕ, καθώς επίσης και με ΜΚΟ. Στις 14 Μαρτίου, Δευτέρα, είχαμε μία συνάντηση προετοιμασίας και είχαμε μία συνάντηση με τη Χριστίνα Κοκκινάκης η οποία είναι, επικεφα... οποία είναι επικεφαλής ε, και στη συνέχεια είχαμε ένα ε, γεύμα εργασίας ε, με πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το απόγευμα είχαμε μια διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο των και στη συνέχεια είχαμε μία συνάντηση με την κυρία Λίζακ ε, που είναι η συγγήτρια ε, για ε, τα ζητήματα μειονοτήτων καθώς επίσης και με τον υπεύθυνο για το Ιράν. και ε, η κυρία Βαλενσιάνο είχε διοργάνωσε ένα γεύμα εργασίας για να συζητήσουμε ε, τις δραστηριότητες του Συμβουλίου. Την επόμενη μέρα συναντηθήκαμε με την κυρία Μπάκτσικ από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης ε, συναντηθήκαμε με τον κύριο Φρανσουά Κρεπό ε, υπεύθυνο για τα δικαιώματα των μετανοστών την κυρία Σπινόσα Κάρσες που είναι η μόνιμη αντιπρόσωπος ε, του Ισημερινό και επικεφαλής της ομάδας εργασίας συναντηθήκαμε με τον κύριο Χαραζάκης με τον κύριο Σουίνκ, ε, διευθυντή του, ε, του, Διεθνής, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, καθώς επίσης και με άλλες ΜΚΟ. Πιστεύω ότι δεχθήκαμε πολύ καλής υποδοχής ε, είχαμε ε, χρήσιμες ε, συναντήσεις, ενδιαφέρουσες, πληροφορηθήκαμε αρκετά. Αρκετοί από τους συζητητές δήλωσαν ότι έχουν κάθε διάθεση να συνεργαστούν με την υποεπιτροπή μας και μια καλή συνεργασία μεταξύ της Γενέβης και του Κοινοβουλίου ήταν κάτι που τονίθηκε τον Ιούλιο επικεφαλής ε, κύριος Λίμ θα έρθει στην υποεπιτροπή μας ε, για να ενημερώσει τα μέλη σχετικά ε, με το έργο που κάνουν ενώ στη συνέχεια είχαμε κάποιες ακόμα προτάσεις να στείλουμε μια πρόσκληση ε, στην ε, υπεύθυνη ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Επιτροπής για να μιλήσει στο Κοινοβούλιο ε, καθώς επίσης και την είπα, τον είπα το εκπρόσωπο πάνω στο θέμα και η πρόκληση αυτή θα επισημοποιηθεί και θέλουμε να διοργανώσουμε και μία εκδήλωση για την πέμπτη επέτειο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, επίσης ε, προσκλήθηκε για να έρθει στην υποεπιτροπή. Αυτό προβλημόταν για πέρσι και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πράξουμε. Κλείνοντας, ήταν μια καλή επίσκεψη και αναγκαία. Ο κύριος Ρέντς, ε, συγητής, εξέφρασε απογοήτευση για την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας όμως λόγω έλλειψης χρόνου θα σταματήσω σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κάρσκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία για παρουσίασε την επίσκεψή μας και θα ήθελα να την ευχαριστήσω και θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Γνωρίζω πως ε, πολλοί ειδικοί εισηγητές τόνισαν την στήριξη που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Επιτροπή μας ε, στην αποστολή τους στα καθήκοντά τους και ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όταν μιλάμε για τις συστάσεις ε, και την διοργάνωση περιπέρου αποστολών στη Γενέβη, θα ήθελα να προτείνω κάτι διαφορετικό, να μην περιοριστούμε μόνο στο να συναντήσουμε τους ειδικού ε, εισηγητές ε, και όσους μας ε, στηρίζουν, αλλά να συναντηθούμε και με όσους έχουν κάποιες επιφυλάξεις για τις δραστηριότητές μας. Μιλήσαμε επίσης και για τη διακίνηση ανθρώπων, την εταιρική ευθύνη ευρωπαϊκών εταιριών γνωρίζω πως ε, αρκετά μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξετάζουν τις δραστηριότητες ε, ευρωπαϊκών εταιριών που μπορεί να είναι επιβλαβής. υπάρχει μία ομάδα εργασίας για τους ε, μισθοφόρους και εξετάζουν τις εταιρείες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι Οι εισηγητές, αυτές, ε, οι εισηγητές αυτοί αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης δεν ε, τους βοηθά. Όταν συναντηθήκαμε με τον Αρμόδιο για την Λευκορωσία, είπε ότι η Λευκορωσία σαμποτάριζε το έργο του και παρόμοια είναι η κατάσταση ε, και για την ομάδα εργασία για τους μισθοφόρους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει, λέει, να συναντηθεί με τους εκπροσώπους αυτής της ομάδας εργασίας. Οπότε νομίζω πως καμιά φορά πρέπει να σκεφτόμαστε και τα όσα πρέπει να βελτιωθούν. Δεν είμαστε τέλειοι. Ε, ειδικά όταν μιλάμε για τη συνεργασία με το Συμβούλιο. Σύντομη παρέμβαση κυρία Τσάμπα από την Κομισιόν. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους βουλευτές για την ενδιαφέρουσα αναφορά σας. Πάντοτε μας ενδιαφέρει το τι γίνεται στη Γενέρη και φυσικά η αντιπροσωπεία είναι έτοιμη να διευκολύνει τις επισκέψεις σας όσον αφορά τα αποτελέσματα. Ε, ε, υιοθετήθηκαν όλες οι πρωτοβουλίες της Ένωσης χωρίς ψήφο για την ανεξιθρησκεία, ε, αλλά ήταν σημαντικό να επανέλθουμε στην ενωπημένη θέση για τα δικαιώματα του παιδιού, διότι το ψήφισμα δυστυχώς ψηφίστηκε στην τελευταία Επιτροπή και και συνδέονταν βέβαια με την σημερινή ακρόαση το πρωί όσον αφορά την κατάσταση στη Βόρεια Κορέα εγκρίθηκε με συνένεση. Δεδομένου ότι το με ψηφοφορία, διότι περιλαμβάνεται η ε, εθάρεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ να σκεφτεί την παραπομπή στο διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο, δεδομένου ότι αυτό το ψήφισμα δημιουργεί ένα πάνελ εμπειρογνωμόνων για τη λογοδοσία, όπω συζητήσαμε το πρωί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίση στήριξε σημαντικέ πρωτοβουλίε για το Ιράν. Ο ειδικό ε, εισηγητή ανανεώθηκε για τη Συρία, ανανεώθηκε η Επιτροπή Έρευνα για τον Νότιο Σουδάν. Δεν δημιουργήθηκε ένα νέο μηχανισμό για να εξετάσει την κατάσταση επιτόπου. Αυτές ήταν προτεραιότητες της Ένωσης. Η Κόρχομ ακόμα πρέπει να αξιολογήσει την σύνοδο. Αυτό θα γίνει ε, στις αρχές του Μαΐου. Δεν μπορώ να σας δώσω πλήρη εξολόγηση, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιη ότι θα υπάρξουν προβληματισμοί όσον αφορά την έλλειψη ενότητας της Ένωσης για ένα από τα ψηφίσματα στο σημείο 7 σε σχέση με τις, ε, ε τους επικισμούς του Ισραήλ. Δεύτερον, Σίγουρα πρέπει να συζητήσουμε τις ανησυχίες και τις τάσεις για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαμε 31 ε, αντίθετε τροπολογίε από την Ρωσική Ομοσπονδία, πολύ αρνητική τάση και θα σκεφτούμε δυνατότητε για να το ε, ξεπεράσουμε αυτό. Και τέλο θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να αντιδράσω σύντομα. Φυσικά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ε, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επισκέφθηκε τι Ρυξέλλες 14 και 15 Μαρτίου. Δυστυχώ συνέπεπτε με το δικό σα συντονισμό. Δεν μπορούσαμε να συνεδριάσουμε εδώ με την υποεπιτροπή σα, αλλά είδε πρόεδρο και άλλου εκπροσώπου, όπω την είπατε εκπρόσωπο. Ήταν πολύ καλή συνάντηση με τον κύριο Λαμπρινίδη. Επίση να σας ενημερώσω Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε δε και με την ομάδα ΠΜΣ που ανέφερε η συγγήτρια. Αυτό που ζητούμε δηλαδή ε, να κάνουν οι άλλοι είναι σημαντικό και για μας ε, να συνεργαστούμε σε ειδικέ διαδικασίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέχασα να σας πω ότι η κυρία Τσάμπα προέρχεται από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Τώρα θα περάσουμε στο τελευταίο, στο ίστατο σημείο της συζήτησής μας για την αντιπροσωπεία στην Καμπότζη. Προείδρευε ο συνάδελφος Βάιντεν Χόλτζερ. 30 Μαρτίου με 2 Απριλίου, δύο μέλη ΕΛΚΑ, δύο σοσιαλιστές, Γκερέρο και Ντέιβιτ Μάρτιν, ένας από τους φιλελεύθερους αεροστρεβήσιους και ένα μέλος των Πρασίνων, η κυρία Λοχμπίλερ. Κύριε Χόλσερ, έχετε το λόγο. Έχουμε λίγα λεπτάκια. Χάρη στην εύνοια των διερμηνέων μας που θα μείνουν λίγα παραπάνω λεπτάκια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος η αντιπροσωπεία αυτή έγινε μετά από δύο ψηφίσματα για την Καμπότζη και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η χώρα ήθελε να αναβάλει την επίσκεψη. Τελικά είχαμε πολύ σημαντικούς ε, συνομιλητές, ε, τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Υφυπουργό Εσωτερικών, βουλευτές, ε, συνομιλία με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών, με ΜΚΟ, με τους επιχειρηματίες και με το δικαστήριο των Ερυθρών Χμέρ. Όπου μιλήσαμε και με εκπροσώπους των θυμάτων. Το κλίμα ήταν ανοιχτό, είχαμε ανοιχτές ε, συζητήσεις και η ανακοίνωση, η δήλωση του τύπου νομίζω δεν ε, ωραιοποίησε τα πράγματα, ήταν, είχαμε όμως ε, σημαντικά αποτελέσματα. Η μεγάλη ανησυχία που είχαμε και προέκυψε αμέσω. Είναι κάτι το οποίο είδατε και στο Μπαγκλαντές, μια πολιτικοποίηση, δύο αντίπαλα στρατόπεδα και ο πολιτικός χώρος ε, σημαδεύεται από αυτό το θέμα και έχουμε βεβαίως συνεχώς περιορισμό της πολιτικής σφαίρας. Είχαμε την περίπτωση του γερουσιαστή Χουντσοκούρ που κρατείται. Επίσης ενημερωθήκαμε για εκστρατείες κατά του Καμψούκα και λοιπόν και άλλα προβλήματα. Βλέπουμε λοιπόν πως α, αντιμετωπίζει προβλήματα η αντιπολίτευση ενώπιση των εκλογών. Περιγράψαμε λοιπόν ποια είναι τα ανησυχητικά σημεία. Η δυνατότητα λειτουργίας των ΜΚΟ συρρυκνώνεται συνεχώς και είχαμε βεβαίως μια ανοιχτή η ε, συζήτηση με διαφωνίες με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών μας έλεγε πως η ΜΚΟ κατευθύνεται από το εξωτερικό ανέφερε τον Βλαντιμίρο Πούτιν για τον ρόλο των ΜΚΟ πράγματα που φαίνονται ανησυχητικά υπήρχε μία συζήτηση και με τους συνδικαλιστές Τώρα δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες. Ε, θεωρώ πως είναι σημαντικό να συνεχίσουμε αυτόν τον ε, διάλογο. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Η αντιπροσωπεία νομίζω κάνει πολύ καλή δουλειά και είναι δικτυωμένη με διάφορα κομμάτια της ε, κοινωνίας. Σημασία έχει και η στήριξη της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής ε, με 10 εκατομμύρια ευρώ που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προετοιμάσουμε τις εκλογές. Το πέρα πρέπει να συζητήσουμε το εάν ε, οι δημοτικές εκλογές οι οποίες αποτελούν, θα έλεγα, πρόβα των γενικών εκλογών, θα μπορούσε να αποτελέσουν αντικείμενο παρατήρησης. Για να δούμε, όπως είπα, τι θα κάνουμε με το μικρό περιθώριο δράσης των ΜΚΟ και όσον αφορά το εργατικό δίκαιο θα πρέπει να δούμε τι γίνεται γιατί η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εντέρος της Καμπότζης η οποία εξάγει φάσματα και ο μεγαλύτερος δωρητής ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρέπει όμως κυρίως να δούμε το ρόλο της αντιπολίτευσης, αντιπολίτευση η οποία δυσκολεύεται πάρα πολύ να παίξει τον ρόλο της ε, και είναι σημαντικό να υπάρχει μια δίκαιη διαδικασία, μια δημοκρατική διαδικασία μέχρι τις ε, εκλογές. Και βεβαίω ε, και αυτοί έχουν αποθέσει τις ελπίδες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να συνεχίσουμε νομίζω αυτές τις επαφές. Δεν ξέρω αν έχουν οι συνάδελφοι κάτι να συμπληρώσουν. Κυρία Στρεβέτσιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, να συμπληρώσω κάποια πράγματα σε αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα κυριότερα ευρήματά μας. Για εμένα η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ε, η κατάσταση της ε, δημοκρατίας στην Καμπότζη μετά τη συνάντησή μας με τα ε, κόμμα εθνικής διάσωσης της ε, Καμπότζης. Ε, δεν έχω καμία αμφιβολία για το ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Έχουμε ήδη τον ίδιο Πρωθυπουργό εδώ και 30 χρόνια. Ο ισχυρός άνδρας της Καμπότζης, ο οποίος ελέγχει ασφυκτικά την εξουσία και τις εξελίξεις στη χώρα και μάλιστα όλες οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για εκφοβισμό και παρενόχληση του κόμματος εθνικής ε, σωτηρίας ε, είναι γνωστές. Μας είπαν ε, πραγματικές ιστορίες και δεν έχω κάποιο λόγο να μην τους πιστέψω. Γι' αυτό νομίζω πως θα πρέπει να επαγρυπνούμε περισσότερο όσον αφορά την κατάσταση στην Καμπότζη ειδικά ε, για τις εκλογές που πλησιάζουν και μάλιστα ε, ίσως θα μπορούσαμε να αποστείλουμε και μία επιστολή στην Βουλή της χώρας δεν πρέπει να μας ξεγελάει να μας ξεγελάνε τα κούφια λόγια που συχνά μας λένε και είχαμε μακροσκελέστατες ε, συναντήσεις αλλά δεν λάβαμε ακριβείς απαντήσεις και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλος δωρητής στην Καμπότζη και μας χρειάζονται και θα έπρεπε να σκεφτούμε μήπως ε, θα έπρεπε η βοήθειά μας να είναι υπόρους. Αυτά είχα και εγώ να προσθέσω. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λοχμπίλερ, τελευταία. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να πω πόσο νομίζω ότι είμαι υπέρ του να απευθύνουμε μια επιστολή στην ε, Βουλή της Καμπότζης και στη Μογκερίνη για να πούμε πως ε, η εμπλοκή μας ε, θα πρέπει να συνοδεύεται από ξεκάθαρα μηνύματα στους εταίρους μας, ειδικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επισκεφτήκαμε διάφορα έργα που χρηματοδοτεί η IDHR και ένα μάλιστα αφορά τις ε, εξώσεις και μάλιστα μας είπαν πως θα δεχτούν αν τους εξασφαλίσουν ε, ε, αξιοπρεπή στέγαση και σχολεία και πρόσβαση στην αγορά. Λοιπόν, ε, οι εκπρόσωποι της ε, κυβέρνησης βλέπω δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία αν δεν επικρατεί η άποψή τους, να το πω έτσι ακούσαμε πως ε, δύο βουλευτές ε, δάρισαν μπροστά στη Βουλή χωρίς να ακολουθήσει κάποια έρευνα και όταν έκαναν πορεία οι συνδικαλιστές στα συνδικάτα το Φεβρουάριο είχαμε απειλές ε, και σκοτώθηκε και ένας εργαζόμενος και όταν είχαμε τις προετοιμασίες για τις δημοτικές εκλογές το 2017 μας είπαν πως ίσως υπάρξει κάποια αύξηση της βίας και δεν μπορούν να το αποκλείσουν. Υπάρχουν νομίζω λοιπόν πολλοί λόγοι την προσωπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρακολουθεί την κατάσταση. Όπως είπα, είχαμε πολλές συναντήσεις με υπουργούς και άλλους. Ε, λυπούμε για το ότι δεν συναντηθήκαμε με τους ομολόγους μας της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν ξέρω, ίσως θα μπορούσαμε να προσκαλέσουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής αυτής ε, ε, φέτος ή του χρόνου για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του νόμου περί συνδικαλισμού Σημείωσαμε την πρότασή σας. Τώρα κλείνει η συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πολύ τους διερμηνείς από όλες τις καμπίνες. Επόμενη συνεδρίαση 15 Μαΐου στις 3.